Αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Γιατί είναι κρίμα να καθυστερούμε την ψηφοφορία και να φερούμε χρόνο από τη συνάντηση με τον Επίτροπο Χόγκαν. Άρχεται η συνεδρίαση λοιπόν. Έχουμε σε 16 γλώσσες διερμηνία, δεν έχουμε σε τεχικά εστονικά, φιλανδικά, μαλτέζικα, σλοβενικά και σλοβακικά. Δεν έχουμε σε αυτές τις γλώσσες. Και περνάμε στο σημείο 11 για τον συντελεστή προσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις του κανονισμού 1306 του 2013 για το ημερολογιακό έτος 2015. Αξιότιμη κύριε πρόεδρε. ευτυχώ. Ε, σας ευχαριστώ που μπορούμε να πούμε δύο λόγια. Έχω μία ερώτηση να κάνω, γιατί είμαι καινούργια στο Κοινοβούλιο σχετικά. Οι προσαρμογέ των άμεσων επιδοτήσεων για το 2015, να τις ψηφίσουμε. Τι θα γίνει με τα μέλη του Κοινοβουλίου που είναι ενεργοί αγρότες. Είναι αυτό πρόβλημα να το διευκρινίσουμε. Δεν ξέρω, γιατί είμαι καινούργια στην Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να το διευκρινίσουμε τι γίνεται με τα μέλη που είναι ενεργοί αγρότες. Έχουμε πολλούς ενεργούς αγρότες εδώ στην Επιτροπή. Βλέπετε, ε, Ανδρέας Γιάρ, Καλινόφσκι, βλέπετε όλοι που χαμογελάν. Ο συντελεστής αναπροσαρμογής αφορά το αποθεματικό. Το αποθεματικό εκτάκτα ανάγκης για το 2015, για τις δύσκολες στιγμές. Το αποθεματικό του 2014 δεν το χρησιμοποίησαμε καν. Οπότε το περιεχόμενο του αποθεματικού επέστρεψε στο προϋπολογισμό και καταβλήθηκε στους γεωργούς. Τώρα έχουμε από τον πρώτο πυλώνα κάποιο συντελεστή. Κάποιο συντελεστή και από αυτό γίνονται κάποιε ενισχύσει. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε στι δύσκολε στιγμές ε, να χρησιμοποιήσουμε άλλα δημοσιονομικά κονδύλια και τα κονδύλια του αποθεματικού τα αφήνουμε για μια πραγματικά δύσκολη και απρόβλεπτη στιγμή. Ε, πέρυσι δεν χρησιμοποίησαμε τα κονδύλια του αποθεματικού και, τα, και επέστρεψαν ε, στον προϋπολογισμό. Και φέτος θα ξαναπροβλέψουμε αποθεματικό για πάνω δεχόμενο. Απευχόμενη βέβαια μια τέτοια κατάσταση, μια εκτακτή ανάγκη που θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει το αποθεματικό. Δεν υπάρχει πρόβλημα πάντως με τους ενεργούς γεωργούς, δεν υπάρχει καμία συμβατότητα. Ο κύριος Δεσπού είναι πραγματικά ενεργός γεωργός. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν θεωρώ ότι είμαι ακροκατελημένος, γιατί δεν ε, έχω πλέον από πέρσι τον Ιούνιο ε, αγροτικές εκτάσεις σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κ. Πόσελτ κατά πόσο μπορούσαν να ψηφίσουν στο παρελθόν συνάδελφοι σε άλλες ψηφοφορίες και τελικά βγήκε ότι ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να ψηφίσει αν τον υπόψη τα κριτήρια Ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Το θέμα δεν είναι να αποκλείσω τον οποιοδήποτε από τη σημερινή ψηφοφορία. Μια ερώτηση από, επί της αρχής σας θέτω ως πρόεδρος. στις επενδυτήσεις οι οποίες άμεσα κατευθείαν πάνε σε ενεργούς αγρότες. Κατά οι ψηφοφορίες που έχουν να κάνουν με άμεσες επιδοτήσεις εδώ στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια, μήπως τίθεται θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Δεν έχει να κάνει αυτό τίποτα με τη σημερινή ψηφοφορία ούτε αποτελεί κατηγορία προς τον κύριο Ντέση ή προς οποιοδήποτε άλλον. Είναι μία ερώτηση. Γιατί δεν θα ήταν καλό να μας κατηγορήσουν ότι ψηφίζουμε εδώ μέσα στην Επιτροπή για τις επιδοτήσεις που θα πάρουμε εμείς οι ίδιοι. Ε, ε, ε, θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά παρακαλώ σύντομα. Ο κύριος Άγνη, που επίσης είναι Γιώργος. Uh, uh, θα ήθελα να διαβεβαίωσω εδώ τα μέλη προς τα δεξιά, αγαπητή κυρία. αν θα μπορούσατε να με κοιτάξετε ότι και είμαι και εγώ ενεργός γεωργός και λαμβάνω την ενιαία πληρωμή για τους αγρότες και δεν ψηφίσω στην πρώτη ψηφοφορία εδώ σήμερα. Εντάξει. Κύριε Σάνρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ε, θέλω να εκφράσω την συμπάθειά μου και το σεβασμό μου προς την συνάδελφο που έθεσε την ερώτηση. Να της πω ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει νόημα. Εδώ έχουμε εκλεγεί. Μετά από δημοκρατικές εκλογές. Έχουμε έρθει εδώ άμεσα και έχουμε κάποια σχέση πάντα με τα θέματα τα οποία συζητιώνται. Έχουμε πολιτικές θέσεις και η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα πράγματι δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ, Ιεράν Καρσία και μετά. Συνάδελφο Ντέ. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει απόλυτο δίκιο. Και επιπλέον, με τον κανόνα των τριών, αν έχουμε κάποια, κάποιο πρόβλημα, οι νεότεροι των 40 ετών ε, Επίση θα μπορούσαν να, να λάβουν μέρο στην ψηφοφορία, γιατί κάποια στιγμή αργότερα θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και να δικαιούνται τι άμεσε ενισχύσει. Οπότε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το επιλύσει η νομική υπηρεσία άλλη στιγμή, όχι τώρα πριν την ψηφοφορία. Συμφωνούμε. Ήρθαμε για να ψηφίσουμε με δεδομένες θέσεις, θέσεις που ανταποκρίνονται στους ψηφοφόρους μας που μας τίμησαν με την ψήφο τους πριν από ένα περίπου χρόνο, στις τελευταίες ευρωεκλογέ. Ας μην χρονοτριβούμε, ας μην καθυστερούμε με τη συζήτηση την ψηφοφορία. Εγώ ούτε Γεωργός είμαι, Ούτε κτηνοτρόφος, ούτε έχω καμιά σχέση με γεωργούς. Ο κύριος Δέσο, ο κύριος Ρόντε και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, παρακαλώ. Γεια, είστε Δέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρακαλέσω και συνάδελφο Έγνο να ψηφίσει, τον συνάδελφο Αγνιό να ψηφίσει δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προπολογισμό στο Κοινοβούλιο επειδή είμαστε όλοι ε, εμπλεκόμενοι. Ε, εδώ πρόκειται για τα θέματα των αγροτών και παράλληλα αυτά πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό έχει να κάνει με τα μονομένα αντικρουόμενα συμφέροντα, όχι με μια μεγάλη μάζα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουν όλοι συνάδελφοι και αυτό έχει διευκρινιστεί εδώ και καιρό. Ο κύριος Ρόντε ακολούθησε τη σειρά των ομιλητών όπως ε, τη συνέταξαν οι, οι βοηθοί εδώ. Δεν ήθελα να σας αποκλείσω κύριε Ρόντα, αλλά προηγούντας τη σειρά ο κύριος Ντες. Γι' αυτό δεν σας έδωσα πριν το λόγο. Τώρα είστε η σειρά σας κύριε Ρόντα. Er Θα ήθελα να τονίσω κύριε Πρόεδρε ότι δεν είμαι γεωργός. Αλλά για 18 χρόνια στην πολιτική που δραστηριοποιούμε. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ τέτοιε ανοησίε. Ακούγοντα την συζήτηση αυτή, η πολιτική εξυπηρετεί συμφέροντα. Εμεί εξυπηρετούμε συμφέροντα. Και ω πολιτική δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούμε ή να θεωρούμε ότι ολυπτούμε ως εκτελεστικό όργανο, ως ε, μέρο τη κλειστική εξουσία θεωρούμε μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει μεροληψία. Αλλά εδώ πέρα δεν τίθεται θέμα μεροληψία. Η πολιτική σημαίνει εξυπηρέτηση συμφερόντων. Αυτή είναι, αυτό είναι ο ορισμό. Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ψηφοφορία για τα πάντα εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια βασική αρχή. Είναι η πρώτη πρώτη σελίδα σε κάθε εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να διακυβερνάτε και να διαχειρίζετε ένα κράτο. Διαβάστε λοιπόν αυτά τα εγχειρίδια και μην σπαταλάτε το χρόνο μα. Πρόκειται για νοησίε, πρόκειται για ε, πραγματικά υπερβολέ σκουπίδια. Τι να πω. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φυσικά. Οποιοςδήποτε πολιτικός μπορεί να ψηφίσει εδώ. Τελεία και παύλα. Ε, ε, Σας ευχαριστώ. Bardzo dziękuję, ale panie pośle, niektóre pokazy... Δεν νομίζω ότι τέτοιες χειρονομίες ε, αρμόζουν στην αίθουσα αυτού, αυτή. Παρακαλώ, αποφύγετε τέτοιες χειρονομίες. Ο κύριος Άγνια, τελευταίος ομιλητής στη συζήτηση. As Απαντώντας άμεσα στον Αλμπερντές, θέλει να ψηφίσω ο κύριος Ντες γιατί πιστεύει ότι σαν Γεωργός πρέπει να ψηφίσω. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως. Είμαι μέλος του UKIP και έχουμε μια διαφορετική στάση και γι' αυτό πήρα την απόφαση σήμερα το πρωί ότι δεν θα ψηφίσω για το πρώτο θέμα πέραν τούτου δεν. Περνάμε στην ψηφοφορία αγαπητοί συνάδελφοι και το ζήτημα της αρχής το διαβιβάζουμε στις ε, νομικές υπηρεσίες για να αποφανθεί. Τα κονδύλια αυτά πάντως τώρα θα μεταφερθούν στο αποθεματικό, αν δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστρέψουν στον ε, προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρουση συμφερόντων σε καμία περίπτωση. Στις 27 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση για τη δημοσιονομική πειθαρχία με βάση την οποία κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υποβάλει μηχανισμό ε, για την εφαρμογή δημοσιονομικής ε, πειθαρχίας τουλάχιστον για τη δημιουργία του αποθεματικού εκτάκτου ανάγκη για τη Γεωργία. Και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουμε μέχρι την 30 Ιουνίου του 2015 για να τροποποιήσουν την πρόταση και να ορίσουν το συντελεστή τη δημοσιονομική πειθαρχία. Οπότε, αν δεν υποβληθούν τροπολογίες, είναι δυνατή διεκπαιρέωση και στην πρώτη ανάγνωση. Η ψηφοφορία θα γίνει στο Κοινοβούλιο κατά την ε, Ολομέλεια του Ιουνίου. Εξέπνευσε η προθεσμία για τις τροπολογίες, δεν κατατέθηκαν τροπολογίες, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε για το συντελεστή αναπροσαρμογής. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε παρακαλώ. ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το θέμα του συντελεστού αναπροσαρμογή. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Ζαμίκαν Τέλος ψηφοφορίας. Έχουμε έναν υπεράριθμο του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Διορθώστε το. Εντάξει τώρα. Κυρία Μαγκίνες. Πρόεδρε, να πω στους συναδέλφους του ΕΛΚ ότι θα φύγω από την ψηφοφορία, θα αποχωρήσω αν ε, είναι και βοηθάει αυτό την ψηφοφορία και τους αριθμούς των ψήφων γιατί με περιμένει κάποιος έξω από την αίθουσα. Εντάξει, ψηφίσαμε. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Βλέπετε 37 υπέρ, 3 κατά. Οπότε περνάμε στο σημείο 12, τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις ε, για τους προϋπολογισμούς 2015 και 2016 έγκριση πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Στο πλαίσια τη ε, ετήσια δημοσιονομική διαδικασία, άπαξ το έτο, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ευρωβουλευτή, επιτροπή ή ομάδα μπορούν να υποβάλουν προτάσει για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει, καθώ και προτάσει για παράταση ε, υπαρχών των προγραμμάτων. Ε, κάτι που θα υποβληθεί σε προκατακτική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έγινε, ε, αυτό γίνεται στις αρχές ή στα μέσα Ιουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας μπορούν ε, να ζητήσουν να υποβληθούν τέτοια προγράμματα πιλωτικά προπαρασκευαστικές πράξεις εκ μέρους της ε, Γεωργικής Επιτροπής. Μάλιστα, 20 Μαΐου στις 20 Μαΐου υποβλήθηκε η, τροπολογία, η προθεσμία για τις τροπολογίες. Λάβαμε 8 προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Αυτά τα 8 προγράμματα και δράσεις θα τα ψηφίσουμε για να δούμε κατά πόσο συγκεντρώνουν την έγκριση της ε, Επιτροπής Γεωργίας. Α, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, δεν είναι 8 αλλά 11 αυτές οι προτάσεις. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έχετε το κατάλογο με τα πιλωτικά προγράμματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου πιλωτικού προγράμματος, παρακαλώ. Διανατάσσετε της χειρός, κατά. Εγκρίνεται το πρώτο. Δεύτερο πιλωτικό πρόγραμμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτό. Τρίτο πιλωτικό πρόγραμμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τέταρτο πιλωτικό πρόγραμμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πέμπτο πιλωτικό πρόγραμμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Κατά, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. Έκτο πιλωτικό πρόγραμμα. Υπέρ. Κατά. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για το πιλωτικό πρόγραμμα υπαριθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αν είχαν σηκώσει το χέρι οι σοσιαλιστές, ε, δεν θα χρειάζεται να το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ του προγράμματος 7. Κατά. Εγκρίνεται. Πρόγραμμα 8. Πιλωτικό πρόγραμμα 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτό. Πρόγραμμα 9. Πιλωτικό πρόγραμμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πρόγραμμα 10. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Και τελευταίο πρόγραμμα 11, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται και αυτό. Από τη στιγμή που βλέπω ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ, δεν θα ρωτώ είναι κατά. Μου το επιτρέπετε. Σας ευχαριστώ. Παίρναμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ο κύριος Ρόντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η ομάδα των φιλελευθέρων θα τηρήσει στάση αποχής στις συμβιβαστικές τροπολογίες και θα καταψηφίσει την έκθεση. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε κατά της έκθεσης αλλά γιατί δεν έχουν υπάρξει καθόλου μα καθόλου διαπραγματεύσεις. Εγώ ζητώ από τους συναδέλφους συντονιστές να πούν στους κοιόδης τους και στους εισηγητές τους, όταν ορίζουν τους εισηγητές, ότι είναι υποχρεωμένοι να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, να μπουν σε διαπραγματεύσεις όταν υπάρχει μια έκθεση αυτό είναι το κοινοβούλιο, αυτή είναι η πολιτική. <clears throat> Και σε αυτή την έκθεση, όπως και στην επόμενη, δεν υπήρξαν καθόλου διαπραγματεύσεις. Και είναι μεγάλη ευθύνη του εισηγητή να ζητήσει από τους σκιώδεις να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Και όχι να γράφει ο καθένας μεμονωμένα ε, την ε, έκθεσή του, να ζητάει από τη γραμματεία να εξετάζει τις τροπολογίες και να κάνει τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι θα ήταν σωστό και δίκαιο σαν συντονιστές να υπογραμμίσουμε αυτό το οποίο σας είπα στους εισηγητές μας όταν ορίζουμε εισηγητές στο εσωτερικό της ομάδας. Γιατί κάθε θέμα, κάθε έκθεση πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, είτε είναι έκθεση είτε είναι γνωμοδότηση. Καλώς, ε, το σημειώνουμε, κύριε Ευρωβουλευτά. θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Γιατί είστε και συντονιστέ, Στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών μπορείτε να το θίξετε. Ο κύριος Χόισλινγκ. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πάρα πολύ συχνά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι εισήγητες. Ε, μας παρουσιάζουν συμβιβαστικές προτάσεις ενώ δεν έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Τι είδου συμβιβασμός είναι αυτός. Ο συμβιβασμός δεν πέφτει από τον ουρανό, είναι καρπός διαπραγμάτευσης. Μπορεί να το δεχτεί κάποιος ή να μην το δεχτεί, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να συμμετέχουν όλες οι ομάδες στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ. Το σημειώνουμε. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος Ρόντε. Αλλά ο εισηγητής δεν είναι παρόν και θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό είναι μια γνωμοδότηση η οποία έπρεπε να ακολουθήσει το χρονισμό της Επιτροπής Προϋπολογισμών ο οποίος ήταν ταχύτατος και γι' αυτό για χρονικούς λόγους, για λόγους χρόνου συγγνώμη, ε, δεν στάθηκε ικανός ο εισηγητής να κάνει προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Πάντως ο εισηγητής δεν είναι παρόν σήμερα εδώ και θα μπορέσει να μας εξηγήσει σε μια μελλοντική φάση. Ε, δεν είχε όμως την δυνατότητα να εμπλέξει τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες με καλύτερο τρόπο. Πάντως το θέμα πράγματι πρέπει να το θέσουμε σε επίπεδο συντονιστών. Ευχαριστώ. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία, ε, γιατί όπως είπαμε θα το εξετάσουμε στους συντονιστέ. Και μία πληροφορία. Ε, δεν έχω ολοκληρωθεί η ουγγρική μετάφραση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ουγγρική μετάφραση. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία του σημείου 13, συγγνώμη, την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Φερνάνδε, ο γενικό εισηγητή για τον προπολογισμό. Εμεί έχουμε συντάκτη γνωμοδότηση. Και η οριστικοποίηση της εντολής θα γίνει με την ψηφοφορία της ε, Ολομέλειας τον Ιούλιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Συγγνώμη, ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρώτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την πρώτη τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Έχουμε έναν υπεράριθμο σοσιαλιστή αυτή τη φορά. Εντάξει, το διορθώσαμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η ψηφοφορία, η τροπολογία, συγγνώμη, 1. Δεύτερη τροπολογία, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 5. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 5. Κατά. Απορρίπτεται η 5. Συμβαστική τροπολογία α. Θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία α. Τροπολογία 11 τώρα του κυρίου Καπούτο. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 11 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία Β. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία Β και περνάμε στην τροπολογία 26 του κυρίου Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 29. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 30. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 31. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Εγκρίνεται. 34. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία γάμα σε. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 44. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 52 του κ. Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 53. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 58 υπέρ, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 61 υπέρ, εγκρίνεται. 62 του κυρίου Ταραμπέλα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 63 υπέρ εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά απορρίπτεται. 66 υπέρ εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται Τροπολογία 75. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 75. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ε, με τις τροπολογίες, όπως έχει τροποποιηθεί μάλλον. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όπως είπε η οριστική εντολή για, το, για τις διαπραγματεύσεις θα υιοθετηθεί 22 και 23 θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ε, το θέμα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Περνάμε στο θέμα 14, το εμπόριο των προϊόντων φώκιας. Αρμόδια καθήλυν επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή ΙΜΚΟ. Εμείς ε, συντάξαμε γνωμοδότηση, ο κύριος Βοητσεχόφσκι ήταν ο συντάκτης και του δίνω το λόγο. Ή μάλλον Ποιος θέλει το λόγο. Θέλει κανείς το λόγο. Ο κύριος Φερά. Ναι κύριε Πρόεδρε, μια επεξήγηση ψήφου. Είμαι υπέρ του υπόστασης του είδους. Αλλά το, η άδεια σκηνηγίου είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τα κράτη. Η απαγόρευση του κυνηγίου δεν είναι, απο, απο, είναι αρμοδιότητα ευρωπαϊκή. Δεν πρέπει η Ευρώπη να α, παίρνει τέτοιου είδους μέτρα. Ο κύριο Ρόντε θέλει το λόγο μήπως. Παρακαλώ. Yeah, uh, we have the same problem here. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα εδώ με αυτό το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως. Δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα και πρόκειται για μια γνωμοδότηση η οποία όχι μόνο θα επηρεάσει πάρα πολλούς συμπολίτε, αλλά κοινωνίες ολόκληρες. Είναι πράγματι απαράδεκτο, είναι φρικτό ε, να είμαστε τόσο περιφρονητικοί απέναντι στον κόσμο τον οποίο η ζωή θα επηρεαστεί μέσα από αυτή την χωρίς καμία διαπραγμάτευση γνωμοδότηση. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω από τον εισηγητή να μου πει γιατί δεν ζητήσατε να γίνουν διαπραγματεύσεις, ποιος ο λόγος. Είναι θέμα αρχής. Ευχαριστώ. Θέλει ο κύριος Βοητσεχόφσκι το λόγο. Ευχαριστώ. Η συζήτηση επί της γνωμοδότησης ε, έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Εγώ απουσίαζα γιατί είχα κάποιες απρόβλεπτες ε, υποχρεώσεις και πρέπει να πάω στην πατρίδα μου. Αλλά η συζήτηση έγινε, η παρουσίαση των επιχειρημάτων έγινε, οπότε δεν ευσταθεί ότι δεν έγιναν ε, συζητήσεις. Άλλωστε η γνωμοδότηση αφορά κάποιους περιορισμούς ανθρωπιστικού χαρακτήρα στο εμπόριο προϊόντων φώκιας. Οπότε από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξετάσουμε το πρόβλημα. Ζούμε στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Και η ανθρωπιστική προσέγγιση και για τα θέματα των ζώων είναι σημαντική πρόκληση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε και να συμφωνούμε ε, βάναυσες συμπεριφορές εις βάρος των ζώων. Και γι' αυτό προτείνονται τέτοιοι περιορισμοί στο εμπόριο. Αυτή είναι κατά τη γνώμη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξού και η γνωμοδότηση είναι υπέρ των περιορισμών. Με εξαίρεση βέβαια κάποιες, α, α, κάποιους πληθυσμούς τοπικούς που έχουν ως βιοπορισμό αυτό το εμπόριο, όπως οι Ινουίτες, ε, Σκιμόοι. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, τη βαναυσότητα της του μαζικού κυνηγιού της φτώχειας της, ε, όπως γίνεται σε ορισμένε χώρες. Νομίζω ότι είναι ανθρωπιστική αυτή η προσέγγιση. Και συμφωνώ ότι σε κάθε ψηφοφορία εκφράζουμε τη γνώμη μας, αλλά το θέμα είναι είμαστε υπέρ της ανθρωπιστικής ε, μεταχείρισης ε, των ζώων και έχουμε και το άρθρο 13 της συνθήκης που καλύπτει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Πώς θέλει ο κύριος Ρόντε το λόγο. Τώρα πρέπει να τα πω δανέζικα. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε πρώτον με ένα εισηγητή ο οποίος δεν ήταν καν παρόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης της έκθεσής του, της νομοδότησής του στην αρμόδια επιτροπή. Ήδη αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει μια κάποια έτσι στάση αλαζονία άμα θέλετε. Δεν συζητήσαμε επί της ουσίας και όπως είπα, επαναλαμβάνω, οι κοινωνίες ολόκληρες που αποτελούνται από κυνηγού επηρεάζονται. Κανένας δεν είναι κατά της φροντίδας των ζώων, αλλά να υπογραμμίσω εδώ ότι και η Greenpeace, όπως επίσης και το WWF, δηλώνουν ότι αυτού του είδους ε, η κυνηγητική δραστηριότητα που διεξάγεται στην Γρυλανδία είναι, ε, είναι βιώσιμη οικολογικά και σύμφωνα με το WWF θα μπορούσαμε και να τριπλασιάσουμε ε, το κυνήγι της φώκιας στις κοινωνίες αυτές χωρίς αυτό να δημιουργήσει προβλήματα αηφορίας. Ο εισηγητής πάνω σε αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί, γιατί δεν μπόρεσε να το συζητήσει με τους υπόλοιπους βουλευτές. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς ε, να συντάσσουμε μία έκθεση, να λέμε τι πιστεύουμε και σκοτιστήκαμε τι λένε οι υπόλοιποι. Διότι ε, αν είναι έτσι τα πράγματα τότε εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω. Έκανε λάθος ο εισηγητής, ακολούθησε λάθος δρόμο το θέμα είναι όπως είπα ευαίσθητο και ο ίδιος ο εισηγητής δεν ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ε, δεν έφερε εις πέρα στο κοινοβουλευτικό του καθήκον. Είναι απαράδεκτο και είναι άδικο απέναντι στις κοινωνίες για τις οποίες συζητάμε εδώ σήμερα. Και είναι άδικο επίσης και εις βάρος των ζώων. Καταρχήν ήταν δικαιολογημένη η απουσία. Ε, πέντε συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό καθένα παρακαλώ και στο τέλο θα δώσω το λόγο και στον εισηγητή μα. Μόι, Χάζερκαμ, Καμ ζήτησαν το λόγο. Γιάρ και Χόισλινγκ. Η κυρία Μόι. Ένα λεπτό όμως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Ρόμπε είμαι είναι ότι δεν ε, λάβαμε υπόψη ε, τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε εμείς να στηρίξουμε ένα τέτοιο σύστημα φρικτών ε, ενεργειών εις βάρος των ζώων αυτών βλέποντας το τι κάνει η Γρυλανδία. Είναι σαφές ότι κάποια από τα γεγονότα στα οποία αναφερόμεθα είναι κατά, αντίθετα με το άρθρο 13 και είναι απαράδεκτη βία η οποία ε, επιβάλλεται στα πτωχά αυτά ζώα. Ευχαριστώ κύριε Χάζερκαμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο Ρόντε ότι ο εισηγητής δεν έκανε και δεν εκτέλεσε καλά τα καθήκοντά του είναι μπορεί να συμφωνεί κανεί ή όχι με την δήλωση αυτή αλλά αντικαταστάθηκε και ζήτησε τη βοήθεια ενός ε, εμπειρογνώμονα στην διάρκεια της επεξεργασίας της έκθεσης. Το θέμα δεν είναι αν θα επιτρέψουμε ή όχι το κυνήγι των ζώων αυτών, αλλά το κατά πόσον θα επιτρέψουμε ή όχι το εμπόριο των προϊόντων αυτών. Και σύμφωνο ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα προϊόντα αυτά. Ευχαριστώ, κυρία Καρεμπάχ. Νομίζω ότι είναι γνωστό ποιε είναι οι απόψει μου. Αλλά να πω ότι υπήρχε σωστή εκπροσώπηση στην Επιτροπή. Συζητήσαμε το θέμα αυτό όπως άρμοζε. Μας διαβεβαίωσε ε, ο εισηγητής ότι θα αποτυπωθούν οι απόψει μα στην έκθεση. Ο κ. Ρόντε δεν προσέγγισε ούτε του υπόλοιπου σκιώδε ούτε εμένα. Και εγώ προσωπικά είχαμε εκφράσει την ε, επιθυμία να πετύχουμε συμβιβασμούς. Αυτό δεν το επιθυμούσε ο εισηγητής και νομίζω ότι πρόκειται για μια φυσιολογική νομοθετική διαδικασία. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει τους εισηγητές να κάνουν οποιοδήποτε συμβιβασμό. Πρόεδρε, από δική μου πλευρά είναι πολύ απλή διαδικασία. Σήμερα ε, καλούμαστε να ψηφίσουμε για το κατά πόσον ε, είναι έτοιμο, έτοιμη η έκθεση προς ψηφοφορία. Θέλουμε να βάλουμε λοιπόν ψηφοφορία ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Τα υπόλοιπα τι να κάνουμε. Τι, να κάνουμε τώρα ε, συζήτηση επί του περιεχομένου. Το θέμα είναι αν θα αναβάλουμε την ψηφοφορία ή όχι. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία, γιατί η ΙΜΚΟ, η Καθήλια Αρμόδια Επιτροπή, θα ψηφίσει στις 4 Ιουνίου. Οπότε αν αναβάλουμε την ψηφοφορία σήμερα δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη η γνωμοδότησή μας. Δεύτερον, ε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ε, από τη συζήτηση αυτή θα αντιλήσουμε όλοι τα κατάλληλα συμπεράσματα. Τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα με την γαλλική διερμηνία. Όχι, εντάξει, διορθώθηκε. Οπότε όλοι θα αντιλήσουμε συμπεράσματα από αυτή τη συζήτηση. Και οι συντονιστές και οι, ο εισηγητής και οι σκιώδης Και θα το συζητήσουμε και στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Πάντως, ε, διαμηνύουμε στους ε, εισηγητές ότι θα πρέπει να έχουν ε, με τους και εισηγητές εκτενέστερες διαβουλεύσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε συμβαστικές τροπολογίες. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε συζήτηση, γιατί όλες οι τροπολογίες θα ψηφιστούν ξεχωριστά. Δεν έχουν συνταχθεί συμβαστικέ τροπολογίες, οπότε ο καθένας θα ψηφίσει τις τροπολογίες. Συμβαστικές τροπολογίες, επαναλαμβάνω, δεν έχουν συνταχθεί. Οπότε δεν μπορείτε να παραπονιέστε ότι παραλήφθηκαν κάποιες τροπολογίες, γιατί θα τις ψηφίσουμε όλες ξεχωριστά. Ο εισηγητή μας και πάλι ο κύριος Βοητσεχόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευνηδιάστηκα και εξεπλάγινα από την προσωπική επίθεση του κύριου Ρόντε, γιατί η, δική μου μεθοδολογία επί της γνωμοδότησης αυτής δεν ήταν διαφορετική από άλλες μεθοδολογίες είτε άλλων εισηγητών είτε σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις εκθέσεις. Και ήδη στο παρελθόν, σε ένα ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της ολοσχερούς απαγόρευσης του εμπορίου προϊόντων φώκιας. Και μάλιστα Είχαμε και προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η κυρία Κάτεμπαχ υπέβαλε τροπολογίες. Δεν έχουμε ουσιαστικές διαφορές στις προσεγγίσεις μας. Οπότε δεν έχουμε τις μορφές σας για καταστρατήγηση των διαδικαστικών κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τηρήθηκαν οι κανόνες και κύριε Ρόντε, ένα λεπτό πριν την ψηφοφορία εξανίσταστε και υποβάλλετε αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, έπρεπε να το είχατε κάνει πολύ νωρίτερα. Γιατί αν είχατε διατυπώσει τις ενστάσεις νωρίτερα, θα το είχαμε συζητήσει. Τώρα ξαφνικά την τελευταία στιγμή, ένα λεπτό πριν την ψηφοφορία, τα διατυπώνετε. Δεν ξέρω τι δεν σας αρέσει στη γνωμοδότηση, γιατί φαίνεται ότι οι επικρίσεις σας είναι γενικές και αόριστες, αλλά δεν επισημαίνεται κάτι θεμελιωδό κακό στην ίδια την γνωμοδότηση. Θα δώσω το λόγο και στον κύριο Χόισλινγκ και στον κύριο Ρόντε στο τέλος για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση και επαναλαμβάνω ότι η γνωμοδότηση είναι ιδιαίτερως ευαίσθητη και λεπτή από κοινωνική και ανθρωπιστική άποψη και ιδεοντολογική συγγνώμη. Γι' αυτό και έχει τόσο έντονο χαρακτήρα η συζήτηση. Ε, μία φορά δεν ε, μπόρεσε να είναι παρόν στη συζήτηση ε, ο συντάκτης γνωμοδότης, αλλά είχε λόγο για την απουσία του. Πάντως όλοι αντλούμε τα συμπεράσματά μας από όλα αυτά. Ο κύριος Χόισλινγκ ένα λεπτό και μετά ο κύριος Ρόντε. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Ρόντε ήπια λίγο πολύ καφέ σήμερα το πρωί μου φαίνεται. Δεν είναι δυνατόν ε, να υποτιμάμε έτσι συναδέλφους. Αυτή είναι η διαφορά με την συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο. Αν δεν κάνει και δεν θέλει να κάνει σε συμβιβασμού ο εισηγητή, ε, είναι δική του απόφαση. Θα ήθελα λοιπόν να το συστήσω να κάνει λίγο πίσω, να υποχωρήσει και να χαμηλώσει λίγο του τόνου. Γιατί αν είναι να κάνουμε τέτοιε συζητήσει ε, πριν από κάθε ψηφοφορία έτσι, θα πρέπει να ψηφίσουμε κάθε θέμα τρει φορέ να το βάζουμε στην ημερήσια διάταξη της ψηφοφορία. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Ρόντα, να ακολουθούμε τέτοιε διαδικασίε. Και ο κύριο Ρόντε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μα. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να κάνω προσωπική επίθεση κατά του εισηγητή. Δεν το γνωρίζω. Αυτό στο οποίο επιτίθομαι είναι ο τρόπο εργασία. Έξι χρόνια είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο και ήμουν συντονιστή επί τέσσερα χρόνια. Και ποτέ ξανά πρέπει να σα πω ότι δεν έχω δει τέτοιο θέμα όπου δεν έγιναν καθόλου διαπραγματεύσει. Εγώ ω κοιόδη δεν νομίζω ότι είναι δικό μου καθήκον να κάνω προς διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι καθήκον του εισηγητή και επίσης θα πρέπει να είναι παρόν όταν συζητείτε στην Επιτροπή το θέμα του. Δεν είναι δική μου δουλειά να πάρω τηλέφωνο τον εισηγητή να του ζητήσω πραγματεύση. Αντίθετα θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Είναι θέμα και αρχής και ουσίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή ε, συμφωνούμε επί της ουσίας δεν χρειάζεται συζήτηση. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου δεν είναι καθόλου συμβατό με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πρέπει να συζητάμε τα θέματα για τα οποία είμαστε αρμόδιοι και τα οποία έχουμε αναλάβει. Και εδώ θα επιμείνω. Και κοιτώντα την ομάδα των φιλελευθέρων, αν θέλουμε υποστήριξη από πλευρά των φιλελευθέρων, θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το οτιδήποτε που δεν έχουμε διαπραγματευτεί εμεί. οι ίδιοι. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με μία παρατήρηση. Οι διαπραγματεύσεις είναι απαραίτητες σε περίπτωση που θέλουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ ε, τροπολογίε ή συμβαστικέ προτάσει. Αυτή τη στιγμή, είπαμε, δεν είχαμε συμβαστικέ τροπολογίε. Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά κάθε τροπολογία. Και θα κρίνετε αν θα την εγκρίνετε ή θα τα καταψηφίσετε. Τροπολογία 26. Ο κύριος ε, της κυρίας Ριμπέιρο ήταν. Επαναλαμβάνω, Το 2009 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπέβαλαν πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων ε, φώκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά όμως από επιτυχή προσφυγή κατά του κανονισμού από τον Καναδά και την Ορβηγία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε να επιφέρει κάποιες αλλαγές με βάση τις αποφάσεις του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ. Όπω σα είπα, αρμόδια καθήλια επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή ΙΜΚΟ και εμεί θα συντάξουμε απλώ γνωμοδότηση. Μάλιστα στι 4 Ιουνίου θα ψηφίσει η αρμόδια Επιτροπή ΙΜΚΟ, οπότε ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα για να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή μα στην ψηφοφορία τη 4 η Ιουνίου στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ξεκινούμε την ψηφοφορία. Τροπολογία. Πρώτη. Τροπολογίες 33, 34, 36, 39, 43 και 48 από κοινού. Ποιος είναι υπέρ από κοινού τις τροπολογίες. Κατά απορρίπτονται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Α, όχι, συγγνώμη. Ήταν μαζί με την 4 πίπτη Η τροπολογία 1 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 1. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37-38. Είναι ταυτόσιμες. Από εκείνο τις ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40, 31, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 7 και 8 μαζί. Λάθος τη δείξα σελίδα. Τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 50. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. 5 και 46 μαζί. Ποιο είναι υπέρ των τροπολογιών 5 και 46. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 5 και 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 49 και 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 2. 52. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 52. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Εγκρίνεται. 45 ποιος είναι... Α, όχι, κατα... καταπίπτει. Γιατί εγκρίθηκε 54. Οπότε περάμε στην 55. Ποιος είναι υπέρ. 55. Κατά. Απορρίπτεται. 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 56. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. 57, συγγνώμη. Ή μάλλον πρώτα την 6, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ της 6. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 7 και 8 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 δεν θα την ψηφίσουμε. 21. Ριμπέιρο. Ποιος είναι υπέρ της 21. Κατά. Εγκρίνεται. 16 και 18. Ποιος είναι υπέρ. 16 και 18 υπέρ. Κατά. Κατά τη γνώμη μου απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 16 και 18. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Εγκρίνεται. 10 και 13 μαζί. Α, όχι, καταπίπτουν οι 10 και 13. Πάμε στη 15. Okay. Ε, όχι, διορθώνει η γραμματεία. Πρέπει να ψηφίσουμε 10 και 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά καταπίπτουν, απορρίπτονται μάλλον. Τροπολογία 15. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Καταπίπτει. 23. 23 ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 25, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24. Ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτα για την τροπολογία 25. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία Κάντεμπαχ. Ζήτησα να επιβραδύνετε κάπως το ρυθμό γιατί καθυστερεί κάπω η διερμηνία μερικέ φορέ και δεν είμαι σίγουρη ότι ψηφίζουμε αυτό που μας ζητάτε. Υπάρχει μια υστέρηση χρονική. Καλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Poprawka 25. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογή 24. Otwier... Ε, kto jest 24? 24 επαναλαμβάνω υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 26 έχει αποσύρθει. Ελεκτρονικός έλεγχος για την 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 26 έχει αποσύρθει. Πάμε στην 27. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. Καλώς. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Α, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Μας έμειναν οι τροπολογίες 3 και 30. Ποιος είναι υπέρ της 3 πρώτα. Κατά. Απορρίπτεται. Και τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Σημείο 15 τώρα. Μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων. Και τροπολογία της οδηγίας του 2003. Η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Χαϊτεμα. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Έμβη, ο Πρόεδρος. 232 τροπολογίε έχουν κατατεθεί, αλλά καλύτερα να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μα για να μα τα εξηγήσει καλύτερα. Εν συντομία όμω, παρακαλώ. Είδε σε έλεγε ο κύριο Χαϊταμα. Οπότε, περνάμε στην ψηφοφορία κατευθείαν. Ξεκινάμε από τη συμβαστική τροπολογία 1. Α. Τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1. Ο κύριος Δες Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το ξαναψηφίσουμε γιατί νομίζαμε ότι ψηφίζαμε το πρώτο σημείο αλλά ψηφίζουμε το συμβιβασμό. Τι, τι ψηφίσαμε δεν καταλαβαμε. Ως πρώτη ψηφοφορία έχουμε την ψηφοφορία της συμβαστικής τροπολογίας 1. και είπα ότι θα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τις συμβαστικές τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 1. Δεύτερο τμήμα. Με την προσθήκη του 2025 που αντικαθιστά το 2020. Ποιος είναι υπέρ. Κανονικά ψηφίζουμε, όχι ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αλλά θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την προσθήκη του 2025. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 76 άρχεται η ψηφοφορία για την 76 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 77 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 78. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, 79 και 81 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 80. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 82, 83 και 84 που είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τροπολογία 85, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 80... 88 και 89 μαζί. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 90. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 11. 11. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 91. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 94 και 95. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 96. Υπέρ εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά απορρίπτεται. 98, 99, 100 και 101 από κοινού. Αλλά πρώτα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 97, γιατί το πρώτο είναι ο εισηγητής. Άρχεται η ψηφοφορία για την 97, τέλος ψηφοφορίας. απορρίψατε. Αυτό είχα πει και εγώ. Τροπολογίες 98, 99, 100 και 101 μαζί. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. Τροπολογία 102. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 103. Ποιος είναι υπέρ? Ντόρφμαν. Ήταν η τροπολογία Ντόρφμαν. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Εγκρίνεται. 104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 106 υπέρ εγκρίνεται. Τώρα 13, 107, 108 και 113 από κοινού. Παρακαλώ ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 109. Ή μάλλον 110 και 111. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Τροπολογία 112 τώρα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 113 δεν ψηφίζουμε. 114, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 115, υπέρ, εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά απορρίπτεται 117 υπέρ κατά απορρίπτεται 118 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 118 άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 119 υπέρ κατά απορρίπτεται 120 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 121 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 122, 123 και 124 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 125, α, ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τρεις τροπολογίες 122, 23 και 24, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, όπως είχα πει. 125, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 126, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά απορρίπτεται τέλος το ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την 130 τέλος ψηφοφορίας το είχα πει απορρίπτεται 131 υπέρ κατά απορρίπτεται 132 υπέρ κατά απορρίπτεται 134 υπέρ κατά απορρίπτεται 133 υπέρ κατά απορρίπτεται 133 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας για την 133 απορρίπτεται 135 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ εγκρίνεται 137 υπέρ κατά απορρίπτεται 138 υπέρ κατά απορρίπτεται 139 υπέρ κατά απορρίπτεται 140 και 141 υπέρ εγκρίνονται. 142 υπέρ κατά απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά απορρίπτεται. 144 υπέρ εγκρίνεται. 145-146. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 147 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 148 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 149 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 150 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 151 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Από κοινό τι τροπολογίε 14, 152, 153, 154, ποιο είναι υπέρ, εγκρίνονται. 155, Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 156, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 156, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Εγκρίνεται. 158. Υπέρ. Εγκρίνεται. 159. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Οκ, okay, για την 159 άρχεται η ψηφοφορία. Otwieram głosowanie 159. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 160. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 161. Υπέρ. Εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά απορρίπτεται 167 υπέρ κατά απορρίπτεται 168 υπέρ κατά απορρίπτεται 169 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογίες 15 και 170 υπέρ εγκρίνονται 171 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16 και 175 υπέρ. Εγκρίνονται. 176 και 177 υπέρ κατά απορρίπτονται. Τροπολογία 180 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά της 182 απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 183 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 19 του εισηγητού επίσης. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 178 και 179. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 184 και 185 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 20 του εισηγητού Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 186. Όχι την αφήνουμε. 187. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 188 και 189. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Εναλλακτική συμβαστική τροπολογία 1. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία της εναλλακτική συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Εκατόν 190 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 191 και 192 υπέρ εγκρίνονται ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 191 και 192 άρχισε ψηφοφορία τέλος Εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα τρία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 194 και 195. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος των 194 και 195. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογία 196. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 197. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογίες 200, 201 και 202 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτονται 203 Πρώτο ηλεκτρονικό έλεγχος των 200, 201 και 202. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτονται. 203. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 204. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 205 και 206. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 207. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 208. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται 209 υπέρ κατά απορρίπτεται 210 210 υπέρ κατά απορρίπτεται 211 υπέρ κατά απορρίπτεται 212 υπέρ κατά απορρίπτεται 213 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 214, 15 και 16 από κοινού. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. 217, 218, 219 και 220 μαζί. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. 221 και 222. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. 223 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερη εναλλακτική συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη δεύτερη εναλλακτική συμβαστική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τη δεύτερη εναλλακτική σύμβαση και τροπολογία. 226 ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 227 ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 228 τώρα υπέρ, κατά, 228. Ποιος είναι υπέρ. 228. Κατά. Απορρίπτεται. Δεν θα ψηφίσουμε την επόμενη εναλλακτική και πάμε κατευθείαν στην δεύτερη συμβαστική, συμβαστική τροπολογία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την συμβαστική τροπολογία 2. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, οπότε πάμε στην τροπολογία... Α, ο κύριος Άγγινιο, συγγνώμη. Στην αγγλική μετάφραση μας ζητήθηκε να ψηφίσουμε για τη συμβιβαστική υπαριθμών 3. Ξεπράσαμε, ξεπράσαμε. Όχι, 2-2. Συμβαστική τροπολογία δύο, δύο. συμβαστικη τροπολογια δύο. ισως εγω εκανα λαθος συμβαστικη τροπολογια δύο. δικιο εχετε Την εγκρίναμε όμως. Και πάμε στην τροπολογία 231. Ποιος είναι υπέρ. 231 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 22 και 232. Ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2.33 υπέρ, 23 ε, συγγνώμη, ε, απορρίπτεται, 24 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 25 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, τροπολογία 26 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, τροπολογία 1 του εισηγητού, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κα, εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 34. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ εγκρίνεται. 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Εγκρίνεται. 40, 41, 42. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτονται 43 υπέρ κατά απορρίπτεται 39 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την συμβαστική τροπολογία 3 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψυχοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία, οπότε πάμε στην τροπολογία 5 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 52. Άρχεται ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Υπέρ τη 7. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 59. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 61. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 του εισηγητού. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62 άρχεται ψηφοφορία. 62 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. 63. Εγκρίνεται η 63 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 64. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Με δύο ψήφους διαφορά εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης, όπως έχει τροποποιηθεί, με ηλεκτρονικό τρόπο. Παρακαλώ, άρχιδη ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Μήπως ο εισηγητής θέλει το λόγο. Έχουμε λίγο χρόνο. Παρακαλώ, θέλετε το λόγο κύριε εισηγητά. Όχι. Συγχαρητήρια πάντως. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι γιατί ήταν πραγματικά άρτια η ψηφοφορία. Ήταν πραγματική ικανοποίηση για μένα η διεξαγωγή αυτής της ψηφοφορίας. Μια και ο Επίτροπος θα έρθει στις 11 ακριβώς, έχουμε ένα τεταρτάκι για καφέ. Επειδή μπορεί να έρθει και λίγο νωρίτερα, να είστε ακριβείς μέχρι τις 11 παρα 5 διακοπή. po przerwie. Μετά την διακοπή, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, θα ξεκινήσουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση που την περιμέναμε πώς και πώς με τον Επίτροπο Χόγκαν Καλωσορίζω θερμότατα τον Επίτροπό μας για να ξεκινήσουμε τον διαρθρωμένο διάλογο με βάση το σημείο 1 του τέταρτου παραρτήματος της Συμφωνίας Πλαίσιο για τις σχέσεις Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής, οι Επίτροποι δηλαδή, έχουν κάθε χρόνο διάλογο με τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές με θέμα την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο χρόνο και την προετοιμασία μελλοντικών δράσεων. Με βάση το διάλογο αυτό, κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή συντάσσει μια έκθεση αποτελεσμάτων, την οποία υποβάλλει στη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών. Η διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος Μπούζεκ θα υιοθετήσει συνοπτική έκθεση και θα την υποβάλει στη διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων. Στην οποία, ο πρόεδρος, στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στη συνέχεια, στην Ολομέλεια του Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί αυτό το ψήφισμα. Θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα την ομιλία του Επιτρόπου και κατόπιν θα δώσω το λόγο στους ε, συντονιστές των ομάδων. Μετά θα ξαναδώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει και θα έχουμε και δεύτερο γύρο με τους ε, υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Σας ε, μοιράσαμε και την ε, χθεσινή επιστολή του Επιτρόπου. στην οποία περιλαμβάνονται πολλές πληροφορίες, πολύ διαφωτιστικές και ενημερωτικές, που θα ληφθούν υπόψη και στην σημερινή συζήτηση. Οπότε κηρύσω την έναρξη της συνάντησής ως τον Επίτροπο και του δίνω αμέσως το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ο διαφερμένος διάλογος είναι βασικό χαρακτηριστικό της διοργανικής μας συμφωνίας και μας επιτρέπει να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα στη Γεωργία το σύνολο των επιτρόπων υπό τον πρόεδρο Γιούνκερ εμένει στον διάλογο μαζί σας και στην στενή συνεργασία και με χαρά συμμετέχω και εγώ στην προσπάθεια αυτή. Είχα έρθει τον προηγούμενο Σεπτέμβριο εδώ για πρώτη φορά και είχα πει ότι σκοπεύω να στηρίξω την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γεωργίας Ελπίζω να σας δείξουμε σήμερα ότι το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αρχίσει να αποδίδει. Εξελίσσεται, περνάει ο καιρός, είμαστε στα μέσα του 2015 και είμαι βέβαιος ότι το feedback, η ανταπόκριση και η ενημέρωση από πλευράς των γεωργών ε, είναι κάτι που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εργασίας μας ε, με σωστό ε, τρόπο. Εσείς είσαστε οι εκπρόσωποι άμεσα εκλεγμένοι των γεωργών που ωφελούνται από την κοινή αγροτική πολιτική και με ενδιαφέρον θα ακούσω τα μηνύματα τα οποία θα μας μεταφέρετε σήμερα στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός προγράμματος εργασίας για το 2016 Μπορεί να έχουμε διαφωνίες σε επιμέρους θέματα, αλλά πρέπει να έχουμε βασικό στόχο την πιο αποτελεσματική κοινή αγροτική πολιτική προς όφελος της υπαίθρου και των γεωργών και να καταστήσουμε την γεωργία ε, πραγματικά κοιτίδα δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανταγωνιστικότητας. Να μειώσουμε την γραφειοκρατία και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε περαιτέρω διακανονιστικές ρυθμίσεις. Βασικά εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να σας ακούσω. Ε, θα μου πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη του προγράμματος το 2015 και θα ήθελα επίσης να μου πείτε και τις προτάσεις σας εφόσον έχετε για το τι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω. Έχουν υπάρξει ορισμένες πρωτοβουλίες για συγκεκριμένες χώρες από τότε που έγινε επίτροπος. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πλατφόρμα για περαιτέρω ε, στενότερη συνεργασία. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα επιτρέψουν να συνεργαστούμε λοιπόν και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την πολιτική μας. Εγώ εμένω στα θέματα της απλοποίησης, της απλούστευσης και έχω ανακοινώσει αρκετά μέτρα για να απλουστευτεί η εφαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής ήδη από το 2015. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές σε επίπεδο κατευθυντηρίων γραμμών. Έχουμε επίσης καθορίσει με διαφορετικό τρόπο και τα φωνοδιαγράμματα για την εφαρμογή. Ε, δεν έχω άλλες παρατηρήσεις εισαγωγικέ να κάνω. Νομίζω ότι θα ήταν πιο παραγωγικό και για τα μέλη του Κοινοβουλίου και για μένα τον ίδιο το να ακούσω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Πολύ καλή πρόταση. Καταπληκτική. Θα δώσω πρώτα το λόγο, όπως είπα, στους συντονιστές που εκπροσωπούν τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας κύριε Επίτροπε για το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα στα πλαίσια του διαστομένου διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε απόψεις και επιβεβαιώνω κύριε Επίτροπε ότι πάντα ήσασταν διτεθειμένος να έρθετε εδώ στο Κοινοβούλιο και πραγματικά έχουν αλλάξει κάποια πράγματα προς τη θετική κατεύθυνση σε σχέση με την προηγούμενη θετία. Τα σημεία από πλευράς της ομάδας μου τα οποία θα ήθελα να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν ε, έχετε ευθύνη για την ευρωτική μεταρρύθμιση, πιο πολύ ευθύνη έχουμε εμεί. Αλλά στα πλαίσια τη γεωργική μεταρρύθμιση αυτή αποφασίστηκε και το screening μετά από ένα έτο, όχι μόνο στα μέσα τη θητεία, να γίνεται, να ελέγχεται δηλαδή πώ εφαρμόζεται η πολιτική. Είναι μεγάλη ευκαιρία λοιπόν αυτή μετά από ένα χρόνο εφαρμογή να δούμε ποια είναι τα πολλαπλά προβλήματα μάλλον ποιε είναι οι, τα αποτελέσματα των πολλαπλών ε, δύσκολων αποφάσεων που χρειάστηκε να λεφτούν. Οι υπάλληλοι μας ε, λέγαν και λένε διαρκώς ότι πρέπει να ρωτήσουμε τους πιο υψηλά ειστάμενους Είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση και οι, οι υπάλληλοι σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να περιμένουμε λοιπόν ένα χρόνο σε θέματα εφαρμογή. Θα είχαμε γλιτώσει πολλά προβλήματα. Πού είναι λοιπόν τα θέματα της ε, εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των θεμάτων από πρώτο πυλώνα στο δεύτερο δηλώνα, ανέκυψε πάρα πολύ η και κάτι θα πρέπει να γίνει λοιπόν για να απλοποιηθεί η κατάσταση. Επίσης κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι κατά πόσον είναι τα κράτη-μέλη υπεύθυνα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει κάποια στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ασάφεια σε ό,τι αφορά τους γεωργούς, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις λωρίδες ασφαλείας, τις λωρίδες ασφαλείας στα χωράφια, οι οποίες από ό,τι φαίνεται απαγορεύονται. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για το πρώτο αυτό έτος, κύριε Επιτροπέ, θα πρέπει εδώ με το να δεσμευτούμε και να αποκοινούμε το ελεγκτικό συνέδριο, να δούμε να γίνει διαφορετικός έλεγχος, γιατί φαίνεται ότι οι αγρότες δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα όλα όσα χρειάζονται. Οι τελευταίες αποφάσεις λοιπόν ελέγχθησαν το Μάιο. Είναι δύσκολο σε αυτό το έτος της οδειάς να είναι πλήρης η εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα πρέπει να τηρηθούν άλλα πρότυπα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Και κάτι άλλο κύριε Επίτροπε. Αυτή η αγροτική μεταρρύθμιση, αν θέλουμε να απλοποιηθεί χρειάζονται και κάποια βασικό δίκαιο. Χωρίς βασικό δίκαιο δεν πρέπει να πετύχουμε τίποτα. Πρέπει να συμφωνήσουμε και μπορούμε να συμφωνήσουμε με το κάθε κράτο μέλο ποια θα είναι τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο βασικό δίκαιο για να μην καταρρύψουμε τη συνολική μεταρρύθμιση, αλλά χωρίς ε, βασικό δίκαιο. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και διαφωνεί η ομάδα μου. Δεν έχουμε χρόνο για να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά χρειαζόμαστε σαφεί κατευθυντήριε γραμμέ σε ό,τι αφορά την αλλαγή τη νομοθεσία, γιατί και οι εθνικέ αρχέ είναι πάρα πολύ μπερδεμένε για το πώ θα γίνει η εφαρμογή. Και τελικά εμά ω κοινοβούλιο θα κατηγορήσουν για την περίπλοκη αυτή διαμόρφωση. Θα πρέπει να φροντίσουμε προκειμένου οι γεωργοί να έχουν τη δυνατότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το greening, το πρασίνισμα, να μπορούν να αντιδράσουν με ευελιξία. Δεν μπορούμε φυσικά να εφαρμόσουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά ακριβώ σε όλη την Ευρώπη με τι ίδιε λεπτομέρειε, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν δώσει πολλές προτάσεις για την απλούσταση της μεταρρύθμισης. Θα πρέπει η αγροτική μεταρρύθμιση να γίνει με τέτοιο τρόπο προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν και να τα καταφέρουν και οι αγρότες και οι εθνικές αρχές προκειμένου και η αγροτική μεταρρύθμιση να συμβάλλει στην εφαρμογή των μέτρων για το περιβάλλον. Αλλά όπως έχουμε πράγματα αυτή τη στιγμή, οι αγρότε πολύ απλά αρνούνται να συνεργαστούν. Θα πρέπει να απλουστευτεί η όλη διαδικασία. Προ το παρόν δεν περιορίζω το χρόνο των συντονιστών. Αλλά θα πρέπει να είστε πιο συνοπτικοί. Ο κύριος Δεκάστρο. Grazie, grazie Presidente e grazie Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χόγκαν που είναι μαζί μας για μια ακόμη φορά μιλώντας για το μέλλον της γεωργίας. Ε, κάθε φορά που μιλάτε για απλοποίηση και απογραφτικοποίηση φυσικά θα είμαστε υπέρ ε, της προσπάθειάς σας και θα σας στηρίξουμε. Είμαστε κατά της γραφειοκρατίας έχουμε ψηφίσει και για μια κοινή αγροτική πολιτική πιο πράσινη στα πλαίσια του λεγόμενου greening, του πρασινίσματος. Αλλά ανησυχούμε. Ανησυχούμε γιατί αυτό το πρασίνισμα σε εισαγωγικά θα περιπλέξει διοικητικά τη δουλειά των γεωργών. Όταν μιλάτε για την απλοποίηση, μας αρέσει αυτό, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι αυτή η απλοποίηση θα είναι μόνο σε επίπεδο βασικών πράξεων, βασικού δικαίου, χωρίς την τροποποίηση των πρακτικών στοιχείων των κανονισμών. Κάτι το οποίο αφήνει πολύ λίγα περιθώρια αλλαγής. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αναθεώρηση ε, μέσα, με στόχο μάλλον ε, την απλοποίηση. Θέλουμε μια πιο πράσινη κοινή αγροτική πολιτική αλλά θέλουμε να καταστήσουμε και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις πιο ικανές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς. Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο είμαστε πάρα πολύ ε, ανήσυχοι, είναι το θέμα της απασχόλησης. Ε, βιώνουμε μια περίοδο κρίσης και η γεωργία έχει δώσει ε, περιθώρια εδώ στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης και μέσω της ανταγωνιστικότητας των εσωτερικών αγορών. Θα πρέπει λοιπόν οι προσπάθειες αυτές να ανταμυφθούν και θα πρέπει να έχουμε σαν βασικό στόχο την ικανότητα της γεωργίας να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες αγορές. Εύθραστες αγορές, αλλάζουν συνέχεια οι διακυμάνσεις των τιμών, οι τιμές μάλλον. Ε, είδαμε τι γίνεται, τι έγινε κυρίως στα γαλακτοκομικά. Το θέμα δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις προς τους γεωργούς, το θέμα είναι τα μέσα που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να διαχειριστούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών που θα είναι όλο και περισσότερο το πρόβλημα για τους γεωργούς. Το είπαμε και χθε στην Ολομέλεια, φρούτα και γάλα για τα σχολεία ε, δεν θα πρέπει εδώ το Κοινοβούλιο να χάσει το δικαίωμα στην απόφαση. Στο Συμβούλιο ακολουθεί άλλη κατεύθυνση και σας ζητάμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα μας στηρίξετε για να καταλήξουμε σε ένα καλό κανονισμό. Υπάρχει η πρόταση και ελπίζω να ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη βιολογική γεωργία με την οποία ασχολούμεθα ήδη μέσω του εισηγητή Χάουσλινγκ Νομίζω ότι και εδώ θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο το οποίο σαφώς και θα βελτιώσει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σταματήσω εδώ Επίτροπε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μας βοηθήσετε για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Έτσι να μην περιμένουμε ε, και να μην ε, έχουμε την ενέργειά μας τραμμένη στην παραγωγή νέων νομοθετικών πράξεων. Το θέμα είναι να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες και να πείσουμε ότι η γεωργία έχει ανάγκη από νέες ε, ε, ρυθμίσεις τις οποίες εδώ σας βοηθήσουμε να περάσουν. Ευχαριστώ. Έχουμε και το Γενικό Διευθυντή πλέμπα που συνοδεύει τον Επίτροπο. Θα ήθελα να τον καλωσορίσω και εκείνον. Και να περάσουμε στον επόμενο μας ομιλητή, τον κύριο Νίκολσον. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με όλους όσοι μίλησαν ε, για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ημών και ημών εδώ σήμερα, γιατί όλοι έχουμε τεράστια ευθύνη στην παρούσα χρονική στιγμή ό,τι αφορά τη γεωργία, όχι μόνο στην περιοχή από την οποία προέρχομαι, αλλά σε όλη την Ευρώπη, γιατί είμαι σε τέτοια επιτροπή πάνω από 26 χρόνια και ποτέ δεν θυμάμαι η βιομηχανία του κρέατος, της γαλακτοκομικής παραγωγής, όλων των κλάδων αυτών να είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Όλοι οι τομείς, όλοι οι κλάδοι αυτοί εκ παραλίλου. Υπήρχαν προβλήματα σε μονομένους τομείς στο παρελθόν, ποτέ όμως όλοι παράλληλα. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν από τους τομείς ε, για τους οποίους καταρτίζω έκθεση σήμερα. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, θα συμφωνείτε, που αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους έξι μήνες ε, είναι η κατάσταση και στον γραφειοκομικό τομέα, όπως είπε και η κ. Δικάστρο δεν συμφωνούμε πάντα και φυσικά αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα και της ζωής και της πολιτικής. Δεν ε, συμφωνούμε για το ότι ο γαλακτικομικός κλάδος αντιμετωπίζει κρίση. Παρά όλα αυτά, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνείτε ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις για τον κλάδο αυτό σήμερα. Γιατί πρόκειται για έναν τομέα που βασίζεται πολύ σε οικογενειακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά πολλών ε, τέτοιων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει την κρίση του κλάδου αυτού. Υπήρξαν διάφορες ε, ε, συγκυρίες που προκάλεσαν δεύτερες μείωσης τιμών και πλέον στην επικράτειά μου οι γεωργοί, οι εκμεταλλεύσεις παράγουν κάτω από την πουλούν κατά από την χαμηλή, από την τιμή παραγωγή. Δεν φαίνεται ότι το ρωσικό εμπάργο θα καταργηθεί σύντομα. Και υπάρχει και η βεβαιότητα του α, καθεστώτος τριμήνου. Πείτε μας όμως ε, πώς εκτιμάτε την κατάσταση στον γαλακτοκομικό κλάδο. Πιστεύετε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες και πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να σας αφήσω επίσης, Επίτροπε. Είπατε ότι θέλετε να βελτιώσουμε τα καθήκοντα του παρατηρητηρίου. Αυτό θα επιτρέψει, λέτε, στο παρατηρητήριο να έχει και να συλλέγει και να παράγει πιο ακριβή στοιχεία, δεδομένα ε, και πιο γρήγορα, προκειμένου να μπορούμε να προβλέπουμε τις κρίσεις και να συστήνουμε δράσεις. Εγώ έχω πει στο παρελθόν ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τι κάνει η Νέα Ζηλανδία και τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εμεί στην Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε ηγετικοί σε ό,τι αφορά τον γαλακτοκομικό κλάδο. Δεύτερη ερώτηση, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω υπερβολικά, για τον προπολογισμό. Είπατε ότι αυτό έχει τις ρίζες του στην πρώτη επίσκεψη που κάνετε στην Επιτροπή. 63 δισεκατομμύρια για την ε, κοινή αγροτική πολιτική κτλ. Θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τον προπολογισμό για τα αγροτικά, γιατί αυτό είναι ο πρώτος και η πρώτη και βασική υποστήριξη της κοινωνικής πολιτικής. Και ξέρετε ότι σε καιρούς ε, οικονομικών δυσκολιών όλοι πρέπει να στηρίξουν το ζωνάρι. Αν είχαμε καταργήσει την ενιαία πληρωμή προς τους αγρότες, που θα καταργηθεί φέτος, στο τέλος του χρόνου, και ξέρετε ότι οι αγρότες που ζουν σε περιοχές που έχουμε στερλίνα που και όχι ευρώ, αντιμετωπίζουν μείωση άμεση, 15%. Ναι, εντάξει, μερικοί θα πούνε να μπούμε στο ευρώ, αλλά αυτό δεν ωφελεί καθόλου τον Γιώργο που προσπαθεί να επιβιώσει. Και αυτό πραγματικά θα φέρει σε δυσχερή θέση πολλούς αγρότες στο Ηνωμένο Βασίλειο του επόμενου μήνε. Θα ήθελα κλείνοντα να πω το εξή. Να εκφράσω εκ νέου την ανάγκη και εσεί και εμεί και το ελεκτικό συνέδριο να συνεργαστούμε πολύ στενά για τομεί όπου εφαρμόζονται νέε πολιτικέ. Όπου υπάρχει δυσκολία ερμηνεία των νέων διατάξεων. Να συνεργαστούμε προκειμένου να μην τελικά ζημιωθούν οι αγρότες για κάτι για το οποίο τον ευθύνονται. Εκτός όλων αυτών, λοιπόν, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ και χαίρομαι που τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Αυτό δεν γινόταν στο παρελθόν και ελπίζουμε να λάβετε υπόψη κάποιες από τις απόψεις που εκφράσαμε. Σας ευχαριστώ. Ε, πάντως, ο χρόνο περνάει, γι' αυτό ρίχνετε και καμιά ματιά στο, μικρό, στο χρονόμετρο όταν μιλάτε, γιατί τρέχει ο χρόνο. Ο κύριο Ρόντε. Ρο... Κύριε Ρόντε, ήρθε η σειρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεστε με το Κοινοβούλιο. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Για τους φιλελεύθερους, για την πολιτική μου ομάδα, μια πιο ενιαία εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι βασικό στόχος. Το είπα πριν και το ξαναλέω σήμερα. Θέλουμε καλύτερα συστήματα ελέγχου, μείωση της γραφειοκρατίας, όπως είπατε κι εσείς, απλοποιημένες διαδικασίες και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε αποτυχημένες πολιτικές που απομόνωσαν τους γεωργούς από τις αγορές. Νομίζω ότι ακολουθείτε τον σωστό δρόμο σαν Επιτροπή. Η ομάδα μου λοιπόν, η ομάδα των φιλελευθέρων, είχε ένα σχέδιο ε, πέντε σημείων για τη συγκεκριμένη νομοθετική περίοδο, το οποίο θα ήθελα συνοπτικά να σας παρουσιάσω. Πρώτον θα θέλαμε εσείς να μας προτείνετε τη μείωση κατά 25% της γραφειοκρατίας και τη μεταρρύθμιση των συστημάτων ελέγχου. Δεύτερον, θα θέλαμε να δημιουργηθούν νέες, ένας νέος κατάλογος προτεραιότητας 10 χωρών με ειδικά μέτρα τα επόμενα χρόνια. Τρίτον, θέλουμε να ανακτήσει την έρευνα στον τομέα αυτό και στην κτηνοτροφία, κυρίως ε, την, οποία, την πρωτοπορία που είχε και να την ανακτήσει ξανά. Αυτό θα ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα οδικό χάρτη για μια πιο έλογη χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα και τέλος, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο τόνωσης της γεωργικής οικονομίας στον τομέα της αντιμετώπισης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών, της μείωσης της εξάρτησης από τρίτες χώρες ε, και της διασφάλισης ε, των προμηθειών τροφίμων σε πολυεθνικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι η βασική τομή στους οποίους θα θέλαμε να δράσουμε και φυσικά και εσείς να κάνετε το ίδιο. Ευχαριστώ. Έχουμε ε, και ε, επισκέπτες του κ. Τεκάστρα από τη Συνομοσπονδία των ε, Ιταλών Γεωργών είστε πια καλεσμένοι ολόκληρη επιτροπή ε, και όχι μόνο του κ. Δεκάστρο. Και έχουμε και εκπροσώπους από την ε, Πολωνική Αυτοδιοίκηση. Καλώ ήρθατε κι εσεί. Η κυρία Σένερα έχει το λόγο. Ε, ή ο κύριος Φλάναγαν που την αντικαθιστά. Ναι, δεν είναι εδώ η κυρία Σύντρες και την αντικαθιστώ Καλώς ορίζω τον συμπατριώτη μου. Έναν άνθρωπο που έχω, στον οποίο έχω πέφτει ερωτήματα σε πολλές περιπτώσεις ε, στο δικό μου κοινοβούλιο. Σε κάποιες περιπτώσεις λαμβάνουμε και απαντήσεις. Ελπίζω ότι δηλαδή δεν συμβεί και αυτό σήμερα. Τα πιο πολλά τα οποία συζητάμε σήμερα εστιάζονται στον πρώτο πυλώνα. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στον πυλώνα 2, τα πράγματα περιπλέκονται ε, καταργούνται τα μικρά προγράμματα τα οποία είναι ουδέτερα σε ό,τι αφορά το εισόδημα των αγροτών. Αν ρωτιέμαι λοιπόν ο Επίτροπος τι πιστεύει για το θέμα αυτό, τι σχεδιάζει να κάνει, γιατί φαίνεται ότι η απλούστευση είναι για τους μεγάλους, με τις μεγάλες πληρωμές και τα πράγματα περιπλέκονται όλο και πιο πολύ για αυτούς που περιμένουν ε, πληρωμές από τον πυλώνα 2. Σε ό,τι αφορά μια δήλωση που έγινε από τον προκάτοχό σας και για τις ανησυχίες που εξέφρασε για τη σύγκλωση που θα γίνει φιλοσικής. Οι φόβοι αυτοί έχουν πραγματικά εκπληρωθεί στην Ιρλανδία αφαιρέθηκαν ε, κάποια ευρώ από τους ε, μεγάλους υποτίθεται για να πάρουν κάποια ευρώ οι μικροί. Αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει σύγκληση. Τουλάχιστον όχι με αρκετά γρήγορο ρυθμό. Και έτσι όσοι εξαρτώνται από τις μικρές πληρωμές αυτές πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να τις λάβουν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περίοδου. Τι θα κάνει λοιπόν στην ενδιάμεση αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να δίνουν τα πολλά στους πλούσιους και ψίχουλα στους μικρούς. Υπάρχουν τέτοια σχέδια. Θα γίνει καν ενδιάμεση αναθεώρηση γιατί σε μία διάσκεψη για τη βιωσιμότητα της ε, αγροτικής απασχόλησης δεν ξέρω αν στέκει αυτό, αλλά άκουσα ότι και την ίδια την ενδιάμεση θεώρηση την αμφισβήτησε. Ελπίζω να γίνει πάντως. Ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή φιλικών ε, απόψεων. Ο Χόισλινγκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρόντε που μου έφερε έναν ε, καφέ δυνατό. Σας ευχαριστώ και σας επιτρόπη που είσαστε εδώ σήμερα και που γίνεται διάλογος όπως και με τον προηγούμενο επιτρόπο, τον τονίζω αυτό. Μας αποστρέφεται μία επιστολή. Κρίμα που έφτασε τελευταία στιγμή. Αλλά αυτή η απόγραφη κρατιοποίηση είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά βλέποντας το τι γίνεται, είναι ακριβώς αυτό που φοβόμαστε το greening δηλαδή βρίσκεται στο στόχαστρο των επιθέσεων. Των επιθέσεων λέω γιατί πιστεύω ότι η μείωση της γραφειοκρατίας είναι καλή και η απορρίθμιση της Επιτροπής ουσιαστικά κατευθύνεται κατά των μεταρρυθμίσεων για το περιβάλλον. Και εδώ πέρα σε εμά σε ό,τι αφορά το πρασινισμά. Είπαμε να βρούμε συμβιβασμούς. Έχουμε μεγάλη ελευθερία δώσει στα κράτη-μέλη και στους γεωργούς να διαλέξουν τι προτιμούν. Και αγαπητέ Άλμπερτ Ντες, ε, μου προκαλεί φρίκι όταν μου λέτε κάθε φορά ιστορίες που έχετε ακούσει από αγρότες. Όλοι βγαίνουν και παραπονιούνται και λένε το μακρύ και το κοντό τους. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτή την μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί. Και πιστεύω ότι τα παράπονα για το πρασίνισμα είναι πραγματικά πολύ υπερβολικά. θα πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στα μέτρα αυτά. Οι φήμες ε, για το ότι δεν είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα αυτά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικές. Χρειαζόμαστε τις πληρωμές ε, τις γεωργικές γιατί έχει απόδοση για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δύσκολη λοιπόν η προσέγγιση αυτή που ακολουθείτε, για να το πω προσεκτικά. Αναφέρατε και κάποιο άλλο σημαντικό σημείο, κύριε συνάδελφε, για το τι ανησυχεί τους ε, γεωργούς. Είναι τα συμπεράσματα των διατάξεων που επιβάλαμε, καταργήσαμε τους ποσοστώσεις, ε, πολλοί είχαν ε, πει ότι θα οδηγήσει σε των τιμών και ακριβώς αυτό συνέβη. Δεν έχουμε καμία απάντηση ένας ολόκληρος ε, κλάδος μικρών εκμεταλλευτών βρίσκονται σε ύφεση και δεν έχουμε καμία απάντηση να δώσουμε. και αυτά που περιλαμβάνονται στο πακέτο για το γάλα δεν θεωρώ ότι απαραίτητα θα έχουν μεγάλα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν κατεπηγόντω να δούμε τι γίνεται με την αγορά. Και θα διαπιστώνουμε και βλέπουμε ότι η απορρίθμιση δεν ικανοποιεί του πάντε σε καμία περίπτωση. Χρειάζομαι κανόνε, χρειαζόμαστε επεμβάσει στην αγορά. Εκτό και αν πούμε. Δηλαδή, τι, λέμε να απελευθερώσουμε εντελώ την αγορά και να δώσουμε και κάποιε μικρέ επιδοτήσει και να δούμε πώ θα λειτουργήσει. Ε, μα δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα έτσι. Ε, ούτε μπορούμε να πούμε ότι στηριζόμαστε στην ελπίδα ότι θα βρούμε νέε αγορέ. Δεν το πιστεύω αυτό. Είσαστε πραγματικά ε, υπέρμαχο του TTIP, κύριε Επίτροπε. Μα το πουλάτε ω η μεγάλη ελπίδα για του ευρωπαίους ε, αγρότε. Δεν έχετε διαβάσει όμω τι μελέτε που έχουν να κάνουν με τι συνέπειε για όλους τους τομείς, για παράδειγμα για τον τομέα της παραγωγής του κρέατος. Α μην υποκρινόμαστε ότι το TTIP είναι ένα σύστημα οικονομικής ανάκαμψης της ευρωπαϊκής αγοράς. Εγώ πιστεύω ότι για τους μικρούς, για τις μικρές εκμεταλλεύσεις θα είναι πιο πολύ πρόβλημα. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο έθιξε ο κύριος Ντεκάστρο για την οικολογική γεωργία και για τις νέες διατάξεις. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει το Κοινοβούλιο και τώρα πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σύμβουλο θα πρέπει να πετύχουν συμβιβασμού και συμβιβασμοί για τον οικολογικό κανονισμό. Η προθυμία σύναψη συμβιβασμών από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξαναγγέλθηκε, δεν βλέπω πού είναι. Βλέπω μάλλον δυσκολίε. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε ό,τι αφορά τι ωριακέ τιμέ για τον τομέα τη οικολογική γεωργία. Θα ήθελα να ζητήσω μια κίνηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην υποστηρίζετε κάτι το οποίο δεν υποστηρίζει τελικά ε, η πλειοψηφία. Σα παρακαλώ λοιπόν ένα πνεύμα συμβιβασμού. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Άγγινιου. Ευχαριστώ. Εγώ άκουσα πολύ χιουμοριστικά εκφράσεις από τον Χάουσλινγκ σήμερα το πρωί, περισσότερο από τα τελευταία έξι χρόνια. Καλό μήνυμα είναι αυτό. Καλωσορίζω λοιπόν και τον Επίτροπο. Καταρχάς, μας δώσατε έξι θέματα έτσι ώστε να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα σε σχέση με τις θέσεις σας. Κοιτάξτε, είναι εύκολο για έναν υπάλληλο να κάθεται σε ένα γραφείο και να γράφει οδηγίες, αλλά είναι δύσκολο για το γεωργό να το θέτει σε εφαρμογή. Πάντως το σημείο 3 και το σημείο 6 είναι πολύ ε, ε, θετικά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα. Ο χρονισμός δηλαδή. Η Βρετανική κυβέρνηση εξόδεψε 500.000 λίρες σε ένα ε, πρόγραμμα πληροφορικής το οποίο δεν ε, ε, δούλεψε ποτέ ε, και απαιτείται μια κάποια ταχύτητα στα πλαίσια του φάσματος των συχνοτήτων για να μπορέσει να λειτουργήσει και στις γεωργικές περιοχές. Δεν έχουν τη δυνατότητα οι γεωργοί να το κάνουν αυτό. Και σύν της άλλης ο χρόνος έχει αρχίσει και περνάει. Ε, ταυτόχρονα η κυβέρνηση είπε ότι τελικά τις οδηγίες αυτές θα τις δώσουμε και σε γραπτή μορφή, θα σας στείλουμε ε, έγγραφα και δυστυχώς ε, δεν το έχουμε δει ακόμα. Ε, είναι σαν να μας λένε ότι έφτασε η επιταγή στο ταχυδρομείο αλλά η επιταγή δεν φτάνει ποτέ. Και αυτή οι οποίοι θα έλεγα είναι η μικρή παραγωγή, αυτοί που έχουν μικρές εκτάσεις με πάρα πολλά επιμέρους κομμάτια για χαρτογράφηση και αυτοί ε, ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουν να συνδυάσουν όλες τις προδιαγραφές. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω μια περαιτέρω παράταση. Ε, παράταση θα το ακούσετε και από άλλους, θα το ζητήσουν και άλλοι. Αλλά νομίζω ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να διευκολύνεται την κατάσταση. Θυμίζω ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι στηρίζουν τα προγράμματα αυτά εν πωλής και για την υπόλοιπη Ευρώπη και δεν θα πρέπει να υφίστανται ζημίες για τις καθυστερήσεις ε, οι οποίες δημιουργούνται οι Βρετανοί γεωργοί ενώ οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ωφελούνται από αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πιστεύουμε εμείς ότι μπορούμε με τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο. Και ακούσαμε σήμερα το πρωί διάφορα για τις εκπομπές διοξιδίου. Κοιτάξτε, ε, πράγματι οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν είναι πάρα πολύ επιτυχημένες, ακόμα και στην κτηνοτροφία ανεξαρτήτως κλίμακας. Το θέμα είναι λοιπόν δεν είναι η συναπόφαση ή κάτι άλλο. Πώς να σας το πω, μπερδεύομαι λίγο. Η συμμόρφωση, η διασταυρούμενη συμμόρφωση, η πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό, αυτός ο όρος, αυτό σημαίνει ότι ε, αν εγώ παράγω για τρία χρόνια το κρέας το οποίο παράγω σήμερα, στην ουσία θα μου επιβάλλεται πρόστιμα. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, θέλω εξηγήσεις. Ευχαριστώ. Όπως σας είχα πει και στην αρχή, μετά το γύρο των συντονιστών θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει και θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος με τις ερωτήσεις των υπόλοιπων βουλευτών. Ο κύριος Χόγκαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συντονιστές για το ευρύ φάσμα των επίκαιρων θεμάτων που μας παρουσίασαν. Θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ε, μετά από τις ερωτήσεις του κυρίου Ντές για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτό είχαμε συμφωνήσει. Μετά από ένα χρόνο θα υπάρξει ε, αναθεώρηση του EFA, ε, δηλαδή των οικολογικών στοχευμένων περιοχών. Από ό,τι φαίνεται σε ορισμένες χώρες δεν υπήρξε η σωστή ερμηνεία αυτών των όρων και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ζήτησα από τους υπηρεσίες μου να ελέγξουν τα θέματα των ερμηνειών και της εφαρμογής και προωθήσαμε κάποιες ερμηνείες που θα είναι χρήσιμες σε σχέση με την εφαρμογή του πνεύματος το οποίο είχαμε στο νου μας σαν συνομοθέτες. και στην ουσία έχει υπάρξει παράταση ε, ε, για πρώιμες πληρωμές για το 2015 και για τις καταγραφές στοιχείων. Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις καρτογραφήσεις των περιοχών EFA, των στοχευμένων οικολογικών ε, περιοχών, όπως επίσης και όλων των διαχωριστικών ζωνών, των συστοιχειών δέντρων, των φρακτών κτλ. Επίσης δεχτήκαμε και την πρόταση που είχατε κάνει τα τέσσερα μέτρα για τη ζώνη διαχωρισμού ε, και τα κενά, τα επιτρεπόμενα μέχρι τέσσερα μέτρα, ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις ορθές πρακτικές, την βιοπικιλότητα αλλά και να προστατεύσουμε λίγο και να ελέγξουμε το δημοσιονομικό κομμάτι. Και γι' αυτό ακριβώς είχαμε εισάγει και τέτοιο είδους περιβαλλοντικά ουσιαστικά μέτρα, ε, έτσι ώστε ε, να μην μπορεί κανείς να πάρει έγκριση για τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις ε, αν δεν έχουν υπάρξει ακριβώς αυτά τα περιβαλλοντικά μέτρα. Λοιπόν τα θέματα της ερμηνείας τα οποία έχουν δημιουργηθεί ε, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία με έχουν απασχολήσει, μας έχουν απασχολήσει και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε εμείς να λιώσουμε το πνεύμα. Από τις 20 Μαΐου πήγαμε 15 Ιουνίου. Υπήρξε μία παράταση. Βέβαια κάποιες φωνές λέγουν ότι υπάρχουν έτσι και αλλιώς προβλήματα σε διάφορες χώρες με το σύστημα εντοπισμού και στο Ηνωμένο Βασίλειο και απαιτείται λίγο μεγαλύτερη ευελιξία. Εγώ όμως δεν είμαι σε θέση μόνος μου να πω για το αν μπορούμε να βρούμε περισσότερη ευελιξία. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη με τεχνικά μέτρα για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων το τακύτερο δυνατόν και με τον πιο ευέλικτο δυνατό τρόπο παρά τα προβλήματα στο τομέα της πληροφορικής. Είναι ένας νέος τομέας έτσι κι αλλιώς και είπαμε για τα EFA, για τους τομείς τους οικολογικούς, ότι δεν θα επιβάλλουμε ποινές ή κυρώσεις στους γεωργούς αν υπάρξει καθυστέρηση στην χαρτογράφηση ε, των περιοχών αυτών και ήδη έχουμε εν πάση περιπτώσει εξαίρεση από τις κυρώσεις, απαλλαγή από τις κυρώσεις για το 2016 μέχρι και το 2017. και όταν υπάρχει μια συνολική δήλωση για ένα τμήμα EFA, για ένα τέτοιο τομέα και μπορούμε να δεχθούμε επίσης από τον ίδιο Γεωργό μια άλλη δήλωση για ένα άλλο τμήμα της γεωργικής εκμετάλλευσης παρότι θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ενιαίο. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις λογικές και στον τομέα αυτό. Αυτό το οποίο θέλω λοιπόν εδώ να πω είναι ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με την εφαρμογή της υπάρχουσας πολιτικής και νομίζω ότι και σε επίπεδο πιθανών αλλαγών νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα μέσω της πιο σωστής ερμηνείας των ρυθμίσεων. Η απλούστευση, το είπα πάρα πολλές φορές, είναι στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης Όλες οι πολιτικές ομάδες που άκουσα προσεκτικά έκαναν κάποιες προτάσεις. Ελπίζω να συνεχίσετε να βοηθήσετε. Ε, νομίζω ότι ε, δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε διαφορετικό δρόμο από εσά. Αν υπάρχουν διαφορές πρέπει να γίνει συζήτηση ε, και να συλλέξουμε ακριβώς τις μεμονωμένες απόψεις που υπάρχουν ιδιαίτερα στον τομέα της απλούστευσης. Ένα από τα θέματα που είπε ο Ντεκάστρο αφορά τα θέματα της, ε, των ε, προβλημάτων της ε, διακύμανσης των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Υπάρχουν προβλήματα εδώ και θα συνεχίσουν να υπάρχουν φοβάμαι, ιδιαίτερα στον γαλακτοκομικό τομέα. Υπήρξε μία μείωση κατά 1,8 τον Μάρτιο της συνολικής παραγωγής γαλακτοκομικού προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική μείωση το 2014 είναι κάτι το οποίο δείχνει τις δυνατότητες προσαρμογής στην αγορά. Ε, κανονικά το 2015 οι εκτιμήσεις ε, λέγουν για μία αύξηση 1% σε σχέση με την ε, αντίθετη τάση το 2014. Νομίζω ότι και οι δυνατότητες νέων αγορών, τις οποίες επιδιώκουμε με πάρα πολύ μεγάλο πείσμα, ε, έχουμε εν ε, θα έλεγα, πετύχει. Έχουμε πολλές δυνατότητες στην Άπο Ανατολή, ακόμα και στην Κίνα και έχουμε επίσης κάποιες δυνατότητες για νέες αγορές και σε χώρες όπως το Μεξικό και νομίζω ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε. Όπως είπα, το 73 επίσης της του χείριου κρέατος που πήγαινε, από αυτό που πήγαινε στην Ρωσία πηγαίνει τώρα στις Φιλιππίνες και σε άλλες χώρες της Άπο Ανατολής. Ε, προσπαθούμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερες τιμές για το χείριο κρέας, αλλά νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η αγορά για τα βιολογικά προϊόντα. Αναφέρθηκε ο κύριος Χάουσλιν και ο κύριος Δεκάστρο. Νομίζω ότι συνεργαζόμαστε για να βρούμε κάποιες λύσεις. Έχουμε έρθει σε στενή επαφή με όλους τους κοιόδης ε, εισηγητές για να δούμε αν χρειάζονται αλλαγές και πού πρέπει οι αλλαγές αυτές να γίνουν. Ε, Το Συμβούλιο ελπίζουμε ότι θα καταλήξει σε συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την ε, τοποθέτησή του τον Ιούνιο του Ιουλίου και ελπίζω και εσείς να καταλήξετε σε συμπεράσματα στο των ετών. Αλλά πολλή δουλειά κάναμε από κοινού σε ό,τι αφορά τα βιολογικά προϊόντα και πραγματικά εκτιμώ ε, τα όσα διαβιβάσατε στις υπηρεσίες μου προσπάθως Θα υπάρξει διακύμανση και αστάθεια. Και ένας από τους τομείς σε ό,τι αφορά το γάλα, πέρα από τις δυνατότητες που μας δίνουν οι ΙΠΑ, είναι το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε την αστάθεια από τις επενδύσεις που κάνουν οι αγρότες σε ό,τι αφορά και την ε, ποσοστώσεις. Και το ίδιο ε, ισχύει και για το μεταπητικό κλάδο σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομιδικά. Να βρούμε λοιπόν μια μέση τιμή και αν σε κάποια χρονική στιγμή υπερβεί η τιμή του γαλακτός στη μέση τιμή, να υπάρχει μια εξισορρόπηση με τον τρόπο αυτό. Αυτή είναι η ιδέα που συζητάμε με την ΕΕ στην πρώτη για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε κάποια πρόοδο προκειμένου για τους νέους ε, Καλλιεργητέ και για τις μικρές επιχειρήσεις να μπορέσουμε να δώσουμε μία πιο σταθερή τιμή μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων σε ό,τι αφορά και το κόστος παραγωγής του γάλακτος. Με πιο προγραμματισμένο τρόπο δηλαδή για μια δεκαετία, περίοδο δεκαετίας. Άρα ασχολούμαστε πολύ με το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά και την Τράπεζα Επενδύσεων. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και θα ελπίζουμε να μπορέσουμε να ε, σα αναφέρουμε τι γίνεται σε σχέση με την ΕΤΕΠ, σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία από κοινού αναπτύξαμε. Ελπίζω λοιπόν να έχω να σας αναφέρω κάποια επιτεύγματα. Η αρχή της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αν υπάρχουν στα αγροτικά προγράμματα οι εγγύησει, αυτά τα οικονομικά μέτρα 100 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα σε ένα ταμείο εγγύησης και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 5-6 φορές για διάφορες επενδύσεις που θέλουμε να κάνουμε στον τομέα των γεωργικών και να μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από τα κράτη-μέλη στο πρόγραμμα ανάπτυξη τη υπέτρου και κάποια κρατημέλη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και θέλουμε λοιπόν να το ακολουθήσουμε αυτό. Τώρα, η 15% μείωση στι τιμέ του γάλακτο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και είναι καλό επιχειρήμα αυτό σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρξει και στενάτερη συνεργασία και να υπάρχει και να μην υπάρχονται οι διακοιμάνσεις αυτές οι τιμές που να είναι επιζήμιες για το Ηνωμένο Βασίλειο. Προσβλέπουμε στη συζήτηση αυτή και ξέρουμε ότι η Ένωση των Γεωργών ήταν πολύ ενθουσιώδης στις προτάσεις αυτές που έκανα στον Μπέρμιγχαμ. Πάντα κοιτάμε λοιπόν τι κάνουμε σε ό,τι αφορά τα θέματα προπολογισμού. Αλλά όπως είπατε χρειάζεται εναρμόνιση και τυποποίηση των όσων κάνουμε από κοινού. Και εδώ κοιτάμε όλο και πιο πολύ την, ε, το σκέλος της απόδοσης σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ. Έχουμε τις επενδύσεις, έχουμε τις δαπάνες, αλλά κοιτάμε κατά πόσον επιτυχάνονται και οι στόχοι. Και αν όχι, πώς μπορούμε να πετύχουμε παρόλα αυτά την επιτεύξη των στόχων. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή των δαπανών ανακράτως μέλος. Άρα συνεργαζόμαστε στενά όλες οι αρχές συνεργάζονται δηλαδή με τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη για τις δαπάνες που υπάρχουν. Το καλωσορίζω λοιπόν αυτό γιατί πιστεύω ότι πραγματικά είναι προστιθέμενη αξία και συνεπάγεται στην προστιθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Να ευχαριστήσω. Τον κύριο Ρόντε για το σχέδιο του με τα πέντε σημεία. Στην προηγούμενη μου ζωή μου άρεσαν τέτοια σχέδια ε, πέντε σημείων, ιδιαίτερα για τι εθνικέ εκλογέ. Γιατί ούτω ή άλλω ο κόσμο πάνω από πέντε δεν ξέρει να μετράει. Οπότε με τα πέντε σημεία επικεντρώνεται σε πολύ σημαντικά μηνύματα. Καλύτερα πέντε από ότι δέκα. Ήδη άμα αρχίσουμε και προσθέτουμε 6-7, αρχίζουν τα προβλήματα. Η μείωση της γραφειοκρατίας και οι κυρώσεις, ε, ε, τι γίνεται με τις, τι γίνεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικαίωχοι στα κράτη-μέλη. Φυσικά χρειάζονται κάποιες μεταρρυθμίσεις, όπως είπε και ο κύριος Φλάναγκαν, και να δούμε ε, να καταλήξουμε σε ένα σύστημα δίκαιο για όλους τους αγρότες που θα λαμβάνει υπόψη το μέγεθός τους, την ικανότητά τους και είμαι υπέρα της απλούστευσης και να δούμε πώς την απλούστευση θα λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις συνιστώσεις, ώστε ε, τους μικρούς καλλιεργητές να τους αντιμετωπίσουμε διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι μικροί καλλιεργητές δεν έχουν ούτε οικονομικές ούτε και διοικητικές ε, ικανότητες να διορθώσουν τα πράγματα. Οπότε οι κυρώσεις ε, κατά αναλογία στους μικρούς ε, καλλιεργητές είναι πολύ ε, χαμηλότερες από τους μεγάλους. Είναι υπέρ αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης. Και η σύγκληση. Φυσικά, απότερο σκοπός είναι η πλήρη σύγκληση, αλλά είναι ευθύνη των κρατών μελών. Και θα έχετε την ευκαιρία να το επισημάνετε και στην πατρίδα σας, ε, που είναι και εκείνη μας πατρίδα άλλωστε. Και από ό,τι ξέρω η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που μέχρι το 2019 θα υλοποιήσει την πλήρη σύγκληση. Βέβαια και άλλα κρατημέλη, αν το επιθυμούν, μπορεί να το κάνουν. Από αυτά εξαρτάται. Και αυτό το νόημα έχει η ευελιξία της ΚΑΠ. Δόθηκε ελαστικότητα και διακριτική ευχαίρεια στους νομοθέτες να το κάνουν. Τώρα, αντιβιωτικά ε, σε ό,τι αφορά την συμπερίληψή τους ε, ε, στη, στη γεωρία και την κτηνοτροφία. Αντιβιωτικά ειδικά στην κτηνοτροφία. Θα μεταφέρω στην κυρία Δριοκάητε τα, το σχέδιό σας με τα πέντε σημεία και για το θέμα αυτό, για να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις ε, της Επιτρόπου για το ζήτημα αυτό. Νέες αγορές. Φυσικά το τελευταίο εξάμεινο ε, είχα ήδη δια, περιοδία, θα τη συνεχίσω το επόμενο εξάμεινο, προσπαθώντας διακαώς να βρω νέες διεξόδους και νέες αγορές ε, για τους γεωργούς μας και τα προϊόντα. Και αυτό έχει επειδή φιλελεύθερος, αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρούμε νέες αγορές ε, για διεξόδους των γεωργικών μας προϊόντων. Και φυσικά ε, συζητώ με τον Επίτροπο Μοέδος για τη βιοοικονομία. Έχουμε στενή συνεργασία και αυτά θα τα εξετάσουμε ιδιαίτερα ε, εν ώψη του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Τα θέματα της βιοοικονομίας είναι πολύ σημαντικά και στη Φιλανδία θα έχουμε 2 δισεκατομμύρια επενδύσεις στη δασοκομεία και τη συμβολή της ε, στην Ήπεθρο και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ήπεθρο, προκειμένου να έχουμε προστιθέμενη αξία που είναι η λέξη κλειδί για την αποτελεσματικότητα. Κύριε Φλάνναγκαν, θα ήθελα να διασκεδάσω τις ε, αμφιβολίες σας για το μήπως αυτό που είπα ε, αν ήταν ηρωνικό ή αστείο ότι δεν θα γίνει διάμεση αναθεώρηση. Έχετε βεβαιώ ότι θα γίνει οπωσδήποτε ενδιάμεση αναθεώρηση. Ίσως λίγο αργότερα, γιατί θα χρειαστεί ε, μετά από μια διετία να ξαναδούμε μερικά πράγματα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν ήταν ηρωνικό για ασία το σχόλιο μου. Επίσης, ε, τα περιβαλλοντικά μέτρα έχουν κέρια σημασία στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και δεν θα μειωθούν, κύριε Χόισλινγκ, ε, οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ χωρίς ε, ισχυρά περιβαλλοντικά μέτρα. Όπου και πηγαίνουν υπάρχουν προβλήματα με το νερό. Και όχι μόνο με την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του νερού. Και γι' αυτό το σχέδιο το επιδετικό του Juncker θα λάβει υπόψη και αυτά τα θέματα, τα περιβαλλοντικά και του ύδατος. Γιατί δεν έχουμε ποιοτικά και ποσοτικά καλό νερό, ε, δεν θα έχουμε γονιμότητα και οι πρώτοι ζημιοθέντες θα είναι οι γεωργοί. Δεν έχουμε λοιπόν κοντόφθαλμη προσέγγιση, αλλά μακροπρόθεσμη και μακρόπνοη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά μέτρα. Μακρηγόρησα μήπω. Τώρα για το TTIP. Δεν πρέπει να αποκλείουμε ε, τη Γεωργία από το TTIP ε, και ούτε το TTIP περιορίζεται στη Γεωργία. Το TTIP είναι ευρύτατη συμφωνία. Δεν περιορίζεται μόνο στη Γεωργία. Θέλουμε μια ισορροπημένη και λογική έκβαση. Εμένα με ενδιαφέρουν οι μελέτε, δεν λαμβάνω βέβαια τα πορίσματα όλων των μελετών, γιατί ακούω για πολλές μελέτες, αλλά ε, κύριε Χόσλινγκ, ε, από τη Γερμανία δεν έχω λάβει καμία μελέτη. Στείλτε τη μου εσείς αν θέλετε. Αλλά είναι σημαντικέ οι στρατηγικές ε, αυτές ε, διαπραγματεύσεις για το TIP. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στι ΗΠΑ πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου το παράθυρο ευκαιρία είναι σχετικά μικρό γιατί θα μονοπολίσει την προσοχή, θα μονοπολίσει την προσοχή προεδρικές εκλογές. Οπότε θα είναι πολύ στενή η ευκαιρία, πολύ το στενό το παράθυρο ευκαιρία. Θα πρέπει να δούμε την ουσία του TTIP, αλλά και φυσικά και το χρονοδιάγραμμα, που όμω είναι πιεστικό, όπω σα είπα, λόγω των προεδρικών εκλογών. Κύριε Άγνιου, η ευρυζωνική στρατηγική που ζητάτε για την Ήπεθρο είναι κάτι ιδιαίτερα προσφυλέ και για μας. Υπάρχουν προβλήματα στην Ήπεθρο με την ευρυζωνικότητα. Θέλουμε όμως να συντονίσουμε 50 διαφορετικά προγράμματα για την ευρυζωνικότητα που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και θέλουμε μονοπευθυντική σειρίδα για να εξασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να έχουμε ένα στοχευμένο ε, πρόγραμμα και μία και να αντιδράσουμε, ε, να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα. 10 με 20% των κατοίκων της υπαίθρου να μην έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ. Τώρα, Beef Genomics, ε, πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή που έχουν τα κράτη-μέλη στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα αυτό με περιβαλλοντικό τρόπο για να μειωθεί ε, η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρόγραμμα διαθέσιμο για να μειώνονται οι εκπομπέ στη γεωργία και να έχουμε και καλύτερα συστήματα εκτροφή για του Ευρωπαίου κτηνοτρόφους. Και η πατρίδα μου μάλιστα αυτή τη στιγμή πρόκειται να εισαγάγει ένα τέτοιο πρόγραμμα και θα μπορούσατε ίσως να το χρησιμοποιήσετε ως μοντέλο για να δείτε αν μπορέσει να λειτουργήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πάνω από 20 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο και θέλουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του Επιτρόπου. Οπότε ένα λεπτό καθένας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ε, ε, για την συνεργασία και παρακαλώ μην επαναλαμβάνετε τις ίδιες ερωτήσεις για να μπορέσει και ο Επίτροπος να επικεντρωθεί σε, στις απαντήσεις. Ένα λεπτό καθένας επαναλαβώ. Ο κύριος Βαλκάρσελ ε, ο πρώτος, που είναι και αντιπρόεδρο, άλλωστε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Σα ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ την προηγούμενη Τρίτη. Συζητήσαμε τα θέματα των οποροκυπευτικών λόγω της, ε, του ρωσικού εμπάργου το οποίο έχει επιβληθεί. Για συγκεκριμένα προϊόντα οι προβλέψεις οι οποίες ε, υπήρξαν για την Ισπανία ήταν ε, ε, ελάχιστες και για προϊόντα όπως τα βερίκοκα, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Ο κύριος Σάπς Έφνης όμως μας έδισε ένα θετικό μήνυμα και εξεπλάγινε όλοι γιατί άρχισε να μιλάει επίσης και για τα μήλα και για τα χλάβια. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια αυτής της κατάστασης ε, ήδη και στα πλαίσια της ε, εισοδείας από το προηγούμενο Απρίλιο είναι θετικό που σε περιλαμβάνει επίσης ε, και τα αμύλες τα πυρηνόκαρπα τις ε, προβλέψεις της και γιατί δεν έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι γεωργοί για τις γεωπολιτικές αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπράναν, παρακαλώ, δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να περιοριστείτε. Επίτροπε, δεσμευθήκατε να μεταρρυθμίσετε το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο το 2016 προκειμένου να δούμε τι γίνεται με την ΚΑΠ και την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα το κάνετε αυτό και δεύτερη ερώτηση. Η ετσιλούσια σύστημα σύζευξης, σύνδεσης ε, επιδοτήσεων στα Σαχαρότευλα είχε μια αναπόφευκτη αλλαγή. 21% διακύμανση, 17 εκατομμύρια επιπλέον. Αυτό ασφαλώ θα σημαίνει επιπρόσθετη πίεση στην παραγωγού ζάχαρης που βασίζονται στις εισαγωγέ αυτές. Αναρωτιέμαι κατά πόσον θα δίνετε εντολή στις υπηρεσίες σας ε, για να εξετάσουν κατά πόσον η τελούσια υποστήριξη, η συνδεδεμένη υποστήριξη μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τις ε, τιμές. Ο κύριος Σεράου Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα που αφορά κυρίως τις αζώνες και που προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα του γάλακτος και της αγοράς γάλακτος. Ακούσαμε τις πρωτοβουλίες που ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά προσέξτε τη συνέπειες που θα έχει η νέα συγκυρία για τα εισοδήματα των γαλακτοπαραγωγών στις εξόχως απόμακρες ε, περιοχές ή στις περιοχές με προβλήματα. Ε, και εσείς ε, από νησί κατάγεστε, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ των νησιωτικών περιοχών, γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη η μεταφορά, η, διά, η διαστάση της αγοράς. πρέπει λοιπόν ε, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις μετά το, την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Επίσης, ε, ε, ελπίζω στο νομοθετικό σας πρόγραμμα για το χρόνο θα στηρίξετε και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή τις ορεινές περιοχές που εξαρτώνται αποκλειστικά από την παραγωγή γάλακτος. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν δίκαια για, το, για την εργασία τους. Επίσης, θα πρέπει να αποφευχθούν αθέμητες εμπορικές πρακτικές και αθέμητος ανταγωνισμός σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ευχαριστώ κύριο Καλινόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε μεγάλες ασυμμετρίες και ανισορροπίες ε, στην ε, αλυσίδα της διατροφής μεταξύ παραγωγών, μεσαζόντων, διανομέων. Πώς θα βελτιώσουμε την ισορροπία στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής τροφίμων, ώστε να έχουμε πιο δίκες ε, και ισόρροπες σχέσεις μεταξύ των κρίκων αυτής της αλυσίδας. Έχετε κάποιες πρωτοβουλίες υπόψη. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη που υπερέβησαν τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις θα πρέπει να καταβάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Και υπάρχει και αστάθεια στην αγορά, αλλά αυτό που επηρεάζεται και από το ρωσικό εμπάργο. Μήπως λοιπόν αυτές τις κυρώσεις θα πρέπει να, και το πρόστιμα να τα, υποβα... να τα διαθέσουμε για την ενίσχυση των γεωργών και για τον εξυγχρονισμό του γαλακτοκομικού τομέα. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγιλέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα εν συντομία να σας εκφράσω τις ανησυχίες, ε, τις ανησυχίες μου ε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ισπανία και σε άλλες χώρες ε, για, την, ε, για το συντελεστή αναπροσαρμογής στις ε, προηγούμενες συμφωνίες δεν έλυσε υπόψη, δεν υπόψη αυτά τα ποσοστά για τους βοσκοτόπους. Τώρα είπαμε ότι δεν θα, δεν θα εφαρμοστεί ο συντελεστής αναπροσαρμογής για τις μειώσεις της έκτασης των βοσκοτόπων και αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες. Στις 15 Ιουνίου λίγη προθεσμία, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, οι ερμηνείς που δίνονται είναι πολύ διαφορετικές για την κατάσταση ε, της εφαρμογής ε, της ε, ΚΑΠ στις διάφορες χώρες. Γιατί πολλοί γεωργοί χρειάζονται τη βοήθεια αυτή από τον πρώτο πυλώνα και έχουν γίνει αλλαγές. Κατάλαβα καλά ότι θα δείξετε ευελιξία αυτά τα χρόνια απέναντι στα κράτη-μέλη μέχρι ότου λάβει χώρα η ενδιάμεση αναθεώρηση. Επίσης, για το πυρηνόκαρπα. Ο τομέα των προεκπαιδευτικών, όπω είπε ο κ. Βαλκάρσελ, αντιμετωπίζει τεράστιε δυσκολίε εξαιτία του ρωσικού εμπάργου. Θα ήταν χρήσιμο να υποβληθούν και συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτραπε να ρωτήσω κάτι από τον κλάδο των απορροκυπευτικών, όχι μόνο από την Ολλανδία, αλλά και από την Πολωνία, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία και το ερώτημα έχει να κάνει με τις πολύ ε, κακές τιμές. Τα έκτακτα μέτρα μετά τις, ε, ε, το εμπάργο τον Αύγουστο του, περι, του περσινού έτους. Και αυτά τα μέτρα σταματούν τον Ιούνιο. Από τα 125 εκατομμύρια λοιπόν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε μια θετική απάντηση γιατί μιλάμε για την εξαγωγή και για τα τιμέ που μειώνονται. Ε, θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία αυτά στο εθνικό αποθηματικό γιατί συζητάμε για πάρα πολλούς αγρότες, για πολλά γενικά ζητήματα, αλλά σε αυτό μπορείτε να απαντήσετε άμεσα και σας ξέρω καλά και ελπίζω να μπορέσετε να απαντήσετε με ένα καταφατικό. Με καταφατικά. Κύριε Ράς Γκαρσία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σα μιλήσω για τον προπολογισμό του 2006. Σήμερα ψηφίσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πιλωτικά προγράμματα για το χρόνο και ένα από αυτά, τα υπέβαλα εγώ, το εγκρίναμε μάλιστα σήμερα, αφορά το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση των κρίσεων, ώστε το παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί για, την, για τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Και ζητώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, τι γίνεται με την πρόταση του Επιτρόπου Ανδρουλάκη για την γενίκευση ε, του συστήματος εμπορευματοποίησης ε, των, των μεταλλαγμένων. Οπότε ουσιαστικά επανεθνικοποιείται η απόφαση για τη χρήση των ε, μεταλλαγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με την νομική ασφάλεια σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά. Γιατί αν κάθε κράτο μέλο, κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει και την πολιτική για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η γνώμη σα σε σχέση με την πρόταση του συναδέλφου σα. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα να εστιαστώ στον γαλακτοκομικό κλάδο. Αναφέρατε ότι εξετάσατε δύο συγκεκριμένες ε, δυνατότητες ε, τη της τη ε, ό,τι αφορά τις ευκαιρίες της αγοράς και την συναλλαγματική ισοδημία. Αλλά στην Βόρεια Ιρλανδία η γεωργοί, οι καλλιεργητές εξακολουθούν να παράγουν κατά από την τιμή κόστους. Θα δεσμευτείτε λοιπόν για να αναθεωρήσετε την τιμή παρέμβασης σε ό,τι αφορά τα Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά τις τιμές και προσπαθούμε να καθησυχάσουμε ε, τις εκμεταλλεύσεις σε ό,τι αφορά την επισήμανση της χώρας προέλευση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία και σε ό,τι αφορά την καλύτερη ρυθμίση. Καλώς ορίζουμε τις ε, προσπάθειές σας, αλλά θέλουμε στη Βόρεια Ιρλανδία να υπάρξουν καλύτερε προτάσεις σε ό,τι αφορά τι τροφικέ καλλιέργειες. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, μια άλλη ερώτηση να σα κάνω. Τις τελευταίες εβδομάδες μιλήσαμε πάρα πολύ για το θέμα των, ε, της μεταναστευσής. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, την βοήθεια για την καταπολέμηση, για την ε, αντιμετώπιση της μετανάστευσης, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην φύγουν, να μην φεύγουν και οι άνθρωποι από την χώρα τους. Και σημαντικός λοιπόν είναι ο κλάδος της γεωργίας. Θέλουμε λοιπόν να μας στείλετε μία επιστολή που θα δηλώνει με σαφήνεια ότι καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχει η γεωργική μας πολιτική. Πρόκειται για μία γεωργική πολιτική που επιτρέπει στον κόσμο να μένει στην πατρίδα του και να εργάζεται στα χωράφια του, να μην λερώσουμε τα χέρια μας με αίμα. Θα ήθελα λοιπόν μια σχετική επιστολή από πλευρά σας και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε επαρκή χρόνο να το συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Γιατί δεν είναι δυνατόν τελικά η γεωργική πολιτική δική μας να οδηγεί τους άλλους σε... να φεύγουν από τις πατρίδες τους. Η επόμενη ομιλήτρια, κύριε Επίτροπε, να μας ε, πείτε... Θα ήθελα και εγώ να λάβω αυτά που στείλετε στα κρατημέλη για το greening, γιατί υποστηρίζω αυτό που λέει ο κύριος Δέση, ότι υπάρχουν ε, βασικά προβλήματα και ότι οι εθνικές αρχές ε, είναι σε μεγάλη σύγχυση. Το πακέτο για το γάλα το εξαντλήσαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ξέρω είναι κατά πόσον προβλέπετε επιπρόσθετα μέτρα σε σχέση με το δίκτυο ασφαλείας το οποίο υφίσταται ήδη. Και αν ναι, ποια μέτρα είναι αυτά. Γιατί πιστεύω ότι η αγορά του γάλακτος και το παρατηρητήριο για την αγορά του γάλακτος εξακολουθεί να έχει καθυστέρηση και ανεπάρκεια ως προς τα στοιχεία που δίνει. Πείτε μας λοιπόν πώς γίνεται και πώς ε, εκτελήσετε η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος γιατί έχουμε μεγάλες εκτάσεις πιο πολλές από ποτέ σε οικολογική προστασία και παρά το γεγονός αυτό είναι όλο και πιο μεγάλες οι πιέσεις που δέχονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που παρήχατε πέρυσι στους χαρακτοπαραγωγούς των βαλτικών χωρών. Και να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, για να στηρίξουμε αυτούς τους γαλακτοπαραγωγούς, γιατί αντιμετωπίζουν κρίση και 15 λεπτά για, του ευρώ για ένα λίτρο γάλα είναι απαράδεκτη τιμή που μάλιστα εξακολουθεί να μειώνεται. Είναι μια πρωτοφανή κατάσταση και αν προηγουμένω οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να πουλήσουν τι αγελάδε του. οι επιστήμονε λένε ότι η παραγωγή γάλακτο θα μειωθεί κατά 20%. Πολύ αρνητικό φαινόμενο και από όσο ξέρω οι Λιθουανοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι ήδη σας έστειλαν προτάσεις για το τι καθεστώ θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Θα πρέπει να συνεχιστεί ε, η συνεργασία ώστε να, αυξήσουμε, ε, ε, να μειώσουμε συγγνώμη, το κόστος της παραγωγής. Ευχαριστώ κύριο Ρεμπέγκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ξεκινώντας θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπατε, ότι δηλαδή 17 χώρες ζήτησαν να υπάρξει παράταση της περίοδου κατά εξάμεινο. Εγώ ήμουνα υπέρ της στρατηγικής αυτής, μελλοντικά στραμμένης πολιτικής, αλλά έχω αρχίσει και ανησυχώ για τον ρόλο ε, των νέων γεωργών. τα μέτρα τα οποία ε, υπάρχουν επαρχούν πιστεύετε ή σκέφτεστε και άλλα μέτρα έτσι ώστε να ενθαρρύνετε τους νέους να παραμείνουν στην Ήπεθρο και ίσως να βοηθήσουμε και νέους να μετακινηθούν από αστικές περιοχές σε γεωργικές περιοχές. Ο ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επιτρόπε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δουλειά σα και ε, δυστυχώ να πω ότι και σε και η Απόστολη δεν μπορούν να είναι εδώ πέρα σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω εξ ονόματό του ε, κάτι για την ευημερία των ζώων. Λέτε, λένε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κοινά πρότυπα για την ευημερία των ζώων για διάφορου λόγου, για να υπάρχουν ίσοι όρια ε, όροι ανταγωνισμού, για να αντιμετωπίσετε με το θέμα των αντιβιωτικών και τη ανθεκτικότητα αυτών, γιατί συχνά συνδέονται με την ευημερία των ζώων. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της καλής εκτροφής των ζώων δεν ορίζεται στη νέα νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει νέος και σωστός ορισμός από άλλα νομοθετήματα, όπως για παράδειγμα το νόμο για την ευημερία των ζώων. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρετε κατά πόσο θα μπορούσατε να θέσετε και να κάνετε λειτουργική αυτή τη νομική διάταξη, προτείνοντας νέα νομοθεσία διευκρινιστική για την ευημερία των ζώων όταν θα εκπνεύσει η υφιστάμενη στρατηγική στο τέλος του 2015. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και για αυτά τα οποία μας είπατε. Ο Χάουσλινγκ έφεσε σημαντικά ερωτήματα για το πρότυπο το γεωργικό το οποίο θέλουμε τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, τι χρονοδιάγραμμα έχουμε και τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να δουλέψουμε επί της ουσίας, αν και διαφωνούμε σε επίπεδο λεπτομεριών. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για τα, για τα βιολογικά προϊόντα. Τώρα για το ξυλέλια φαστιδιόζα. Τι γίνεται με τα όρια ελέγχου εισαγωγής φυτικών προϊόντων και πώς εσείς στα πλαίσια του πακέτου για την υγεία να προχωρήσετε και στην προστασία, προστασία των φυτών ε, από τις εισαγωγές επικίνδυνων προϊόντων. Τώρα για το TTIP είπατε σωστά ότι το χρονοδιάγραμμα πηγαίνει αρκετά στο μέλλον. Αλλά έχουμε πάρα πολλές ανησυχίες ιδιαίτερα για το βόλιο κρέας και για το γάλα. Πώς θα διατηρήσουμε τη γαλακτοπαραγωγή στις ορεινές και υπεπεθερικές ζώνες. Ο Γιάρ, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και πέρα από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι να κάνω δύο παρατηρήσει. Καταρχά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βόλιο κρέας. Ήθελα να δω τι θα επιλέξει ο Επιτροπός από τις ε, πολλαπλές ε, ε, προτάσεις, αλλά πιστεύω ότι οι προτάσεις που συζητιώνται είναι μια καλή αρχή. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Κατά δεύτερον, να συνεχίσετε το διάλογο με τους γεωργούς. Αυτό οδηγεί σε νέες διαπιστώσεις. Παρευρεθήκατε στη λειψία και συζητήσατε με τους ε, αγρότες. Το πρώτο λοιπόν συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι ότι ήταν αμφιλεγόμενο στη Γερμανία κατά πόσο θα μπορούσαμε στο Δεκέμβριο να κατατηθούν και να πληρωθούν οι επιδοτήσεις αλλά πραγματικά εκεί κινήσατε κάτι και θα πρέπει να το συνεχίσετε λοιπόν αυτό τη συζήτηση για την μείωση της γραφειοκρατίας. Σας παρακαλώ να συμφωνήσουμε τι έχει νόημα και αν αυτό δεν αγγίζει το βασικό δίκαιο, έχει καλώς. Αν και στην περίπτωση που αυτό θα αφορούσε και το βασικό δίκαιο, να το κοιτάξουμε λοιπόν από κοινού για να συμφωνήσουμε τι θα πρέπει να αλλάξουμε. Ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σας. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Στα πλαίσια μιας πρόσφατης επαφής με έναν Γάλλο υπεύθυνο που ανήκει σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του είχε ζητήσει να αρθεί το εμπάργο για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Τι ακριβώς γίνεται. Δεύτερον, μιλήσατε για το διεθνές εμπόριο. Μπορείτε να μας πείτε αν είμαστε σε θέση εμείς να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που δημιουργούνται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής που κάθε φορά που έρχονται στο Κοινοβούλιο μας ζητούν να υπάρξει μια συμφωνία ανταλλαγής ενέργειας με τρόφιμα. Η υπηρεσία σας έχουν αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα. κύριε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, προηγουμένω ε, μιλήσατε για τη σύγκληση και είπατε ότι είναι καθήκον των κρατών μελών. Φυσικά εδώ από νομική άποψη έχετε δίκιο, αλλά να μην απαλλαχτείτε και από τη δική σα ευθύνη. Η μεταρρυθμίση η οποία εφαρμόζουμε ε, δημιούργησε τις ε, συνθήκε με τι οποίε μια χώρα όπω η δική μου η Ιταλία να υπάρχει πλέον αναλογία μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα ε, ένα προς 10. Δηλαδή, ε, σε εμάς ένας αγρότης μπορεί να παίρνει 50 ευρώ, ενώ μερικά χιλιόμετρα παραδίπλα ο ανταγωνιστής του να παίρνει 500 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το στοιχείο αυτό και στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Τι γίνεται με την κατανομή του πρώτου και κατά πόσο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις. Ευχαριστώ. κυρία Ζουφίρα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, Επίτροπε, η οποία είναι πράγματι πάρα πολύ χρήσιμη. Θα ήθελα να αναφερθώ στα βιολογικά προϊόντα που είναι ένας τομέας που αυξάνεται συνεχώς. Ξέρετε ότι αυξάνεται ε, η κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων όπως και οι γεωργικές εκτάσεις που τα παράγουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες απορίες όμως και φόβοι στους γεωργούς ε, για να επενδύσουν στον τομέα αυτό γιατί δεν ξέρουν πώς θα μπορέσουν να αλλάξουν αυτούς τους κανόνες. Δεν υπάρχει αμφιβολία όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Αντρέο ότι υπάρχει ανάγκη από ξεκάθαρους κανόνες και θα πρέπει να έχουμε σωστές επενδυτικές κατευθύνσεις. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας γι' αυτό και θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε για τα μέτρα τα οποία θα προβλέψει ο νέος αυτός κανονισμός σε σχέση με το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. κύριος Συνέκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα μιλήσω για το TTIP. Η γεωργία είναι μόνο το 5% της ε, διαδικασίας ε, των διαπραγματεύσεων του TTIP. Και ε, έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία των διαφορών κλάδων. Και τα, η αγροτική τελωνιακή δασμή είναι 6,6% στις Ηνωμένες Πολιτείες και 12,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στις αυστηρότερες ε, νομοθετικές διατάξεις που έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και φθηνότερη ενέργεια και φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει κάποια πιθανότητα να αρθούν ε, οι δασμολογικοί φραγμοί. Υπάρχει καμιά πιθανότητα να παραμείνουν οι προδιαγραφές ε, ε, όπως έχουν, δηλαδή χαμηλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυστηρότερες ή ψηλότερες για μας, γιατί έτσι επιδεινώνουμε τη θέση των γεωργών μας. Επίσης, οι γεωργοί στην Βουλγαρία προσβλέπουν στη συνάντηση μαζί σας στην ετήσια γεωργική έκθεση. Θα είστε πρόσδεκτος κύριε Επιτροπέκη. Ο κύριος Βοητσεχόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Πολωνία έχουμε νέο πρόεδρο, τον συνάδελφο Ευρωβουλευτή Άντζεϊ Ντούντα και στις τελευταίες μέρες της προεκλογικής της ε, επισκεφθήκαμε Αγροτικέ εκμεταλλεύσει, ε, κτηνοτροφικέ συγκεκριμένα μονάδες και ωραίες ε, αγελάδες, ε, συνάντησε ο κύριος Ντούντα, αλλά ήταν θλιβερό το αποτέλεσμα γιατί ο κτηνοτρόφος, ο του είπε ότι θα πρέπει να πουλήσει το κοπάδι του γιατί δεν είναι πια βιώσιμη η παραγωγή γάλακτος εξαιτία των χαμηλών τιμών και των μεγάλων εμποδίων που υπάρχουν. Οπότε θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Καρινόφσκι και άλλοι συνάδελφοι και να σας ζητήσω, ε, κύριε Επίτροπε, να δούμε τι θα γίνει με τις κυρώσεις. Βέβαια δεν επαφίεται αυτή η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά στο Συμβούλιο. Αλλά σε περίπτωση που έχουν καταργηθεί οι ποσοστώσει, ε, δεν έχει νόημα να πληρώνονται αυτέ ε, οι κυρώσει και τα τεράστια πρόστιμα από του γεωργού πολλών χωρών μελών. Και μάλιστα είναι αδικαιολόγητη αυτή η επιβολή κυρώσεων. Από τη στιγμή που καταργούμε τις ποσοστώσεις, γιατί να παραμένουν ενισχύ οι κυρώσεις που δημιουργούν τεράστιες απειλές για την επιβίωση των γαλακτοπαραγωγών Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Ελάχιστο χρόνο έχουμε ακόμη. Θα παραμείνουν λίγο μαζί μας ακόμη οι διερμηνείς επαναλαμβάνουμε τα προβλήματα της ε, γαλακτοκομικής ε, παραγωγής που είναι συγκυριακή ή θα παραμείνει. Ε, θα πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις και πώς θα διορθώσουμε αυτή την κρίση. Σε ό,τι αφορά το TTIP. Το TTIP δεν αφορά φυσικά μόνο τη γεωργία. Αλλά όλο και πιο συχνά στις διεθνείς συμφωνίες πολλά πράγματα συμφωνούνται ερήμην ή πίσω από την πλάτη των γεωργών και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά χαιρόμαστε ιδιαίτερω ε, για αυτά που μας είπατε ότι θα ανασταλούν ε, οι κυρώσει προς τους γαλακτοπαραγωγού. Αυτή είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Και επίση στο μέλλον θα πρέπει ε, να παρακολουθούμε καλύτερα την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να κάνουμε και αυτή την αναθεώρηση. Επίσης, ε, θα έχουμε αρκετό χρόνο για να υιοθετήσουμε αυτές τα, αυτά τα μέτρα και θα τα δουν οι γεωργοί ή θα έχουν κλείσει στο μεταξύ της δραστηριότητας τους, όπως είπε ο κύριος Χόισλινγκ. Ε, πάντως, εμείς ε, σας νιώθουμε σαν το δικό μας επίτροπο και δεν μπορούμε αυτό να το πούμε για κανέναν άλλο επίτροπο. Σας ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο. Thank you very much, Chairman. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρκετοί αναφέρθηκαν στα οπροκυπευτικά και στο ρωσικό εμπάργκο. Γνωρίζετε ότι εγώ έχω επεκτείνει το χρόνο για τα μέτρα τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από τον προηγούμενο Αύγουστο. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα που επηρεάζονται. Αρκετές χώρες ε, έχουν ε, κάνει όμως και διάφορες αναφορές για προϊόντα που δεν έχουν σχέση με το ρωσικό εμπάργο. Ε, θα πρέπει να δούμε ε, τι προϊόντα υπάρχουν και είδαμε τι γίνεται με τα πυρηνόκαρπα. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει οι αιτήσει των κρατών μελών να έχουν σχέση με προϊόντα που επηρεάζονται από το ρωσικό εμπάργο και μόνο. Η μεταρρύθμιση ή μάλλον η επανεξέταση η οποία θα γίνει το 2016 ε, νομίζω ότι έχουμε μια κάποια έλλειψη χρόνου και έχω την εντύπωση ότι θα ξεκινήσουμε λοιπόν στις αρχές του 2016 την επανεξέταση των μέτρων. Τώρα, δημιουργήθηκε και μια ειδική ομάδα σε σχέση με το καθεστώς της ζάχαρης και την κατάληξη του προγράμματος στο τέλος του 2016. Να σας θυμίσω ότι η εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη, συμμόρφωση, στήριξη μάλλον, ε, έχει σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία υφίστανται πιέσεις ή με συγκεκριμένες κατηγορίες των γεωργών και τα κράτη-μέλη είναι αυτά που κάνουν τις προτάσεις. Για τις αζόρες τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το 27% του, ε, της αγοράς γάλακτος προέρχεται από τις αζόρες. Έχουν επίσης ε, υπάρξει πολλές δυνατότητες ε, για επενδύσεις στους γεωργούς. 125 ευρώ ανά η Ελλάδα έχουν επίσης ε, δοθεί προς τις Αζόρες περισσότερο από ό,τι στην Μητροπολιτική Πορτογαλία. Νομίζω ότι αυτά τα μπόνους, τα μπόνους τα οποία μπορεί να πάρετε για το προϊόν σας είναι ένα πολύ καλό και γενναιόδωρο και νομίζω ότι και σε σχέση ε, με τα επιμέρους μέτρα της περιφερειακής κυβέρνησης θα μπορέσετε να καλύψετε τις ανάγκες ε, των, ε, των κτηνοτρόφων και των γαλακτόπαραγωγών. Ε, απαιτούνται τέτοια μέτρα για να ισορροπήσει η αγορά στον χαλακτοκομικό τομέα. Κατανοώ ότι όλοι θέλουν περισσότερα, αλλά το πρόγραμμα θα αναθεωρηθεί στα τέλος του 2016 και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές έτσι ώστε να βοηθηθούν ε, και η παραγωγή των αζωρών αλλά και άλλων νήσων που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Ε, πολλά ακούστηκαν επίσης για τις ορεινές περιοχές και συμπληρωματική στήριξη. Αυτός είναι ο ρόλος των ε, προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου. Εκεί τα Υπουργεία σας πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουν τώρα. Δεν είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, απαιτούνται όμως συγκεκριμένα προγράμματα για τις απομεμακρυσμένες περιοχές και τις ορεινές περιοχές που χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Λοιπόν, οι συνδεδεμένες αυτές μορφές λοιπόν στήριξης πρέπει να απευθυνθούν και να τις ε, φέρει πέρα σε εθνικό επίπεδο κάθε χώρα. Οι γεωργοί θα πρέπει να πάρουν ε, πάνω από το ποσοστό το οποίο τώρα τους ανήκει στα πλαίσια της αλυσίδας ε, της διατροφικής Μιλήσαμε και με την κυρία Χάουσκε και είδαμε πώς η αντίστοιχη γενική διεύθυνση θα μπορέσει να κάνει προτάσεις που να βοηθήσουν τους παραγωγούς οι οποίοι ίσως το τελευταίο καιρό έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της πίεσης την οποία υφίστανται από τους άλλους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αυτή. Λοιπόν, οι αρμόδιες Ευρωπα... οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν το θέμα και θα μπορέσουμε εμείς να βρούμε περαιτέρω τεκμήρια έτσι ώστε ε, να μην μειώνεται η αποδοτικότητα της γεωργικής δραστηριότητας από την υπερβολική πίεση των υπολείπων συμμετεχόντων στην διατροφική αλυσίδα. Νομίζω ότι και για την Ισπανία Μιλήσατε και για την... Ε, We've made in the changes in recent times is interpretation. Η συνδεδεμένη στήριξη επίσης νομίζω ότι η πλήρη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών θα ήταν κάτι το θετικό για τους γεωργούς. Αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ εγώ ότι θα γίνουν ε, περισσότερες αλλαγές, μίζωνες αλλαγές, παρά στο επίπεδο της ερμηνείας μόνο των κανόνων αυτών στα πλαίσια της απλοποίησης της εφαρμογής των μέτρων μας σε εθνικό επίπεδο και όπως είπε και ο συνάδελφός σας και εσείς θα επανεξετάσουμε το θέμα των πυρηνοκάρπων. Αναφερθήκατε και στις, στον, ε, συνέπειες του ρωσικού εμπάρκου στις τιμές. Θα δούμε τι γίνεται μέχρι το τέλειο Ιουνίου για να αναθεωρήσουμε την κατάσταση, τι γίνεται με τα φρούτα και μετά τη στήριξη που δώσαμε στον τομέα των απορροκυπευτικών. Αλλά ε, είπατε, μιλήσατε γενικά για τις τιμές, δεν νομίζω το σχολείο σας αφορούσε ιδιαίτερα το ρωσικό εμπάργο. Πρόκειται για μια πολιτική που προσανατολίζεται προς την αγορά και αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε και ε, υιοθετούμε και μέτρα πρόθεση για την αναζήτηση νέων αγορών. Έχουμε σημαντικό προπολογισμό για την ε, προβολή και την πρόθεση των προϊόντων στα πλαίσια της ΚΑΠ για την επόμενη διετία. Δεν έχουμε ε, πάντως ε, άμεσα σχέδια για παρέμβαση στην αγορά προϊόντων και ιδιαίτερα στα απορροκυπευτικά. Τώρα, μιλήσατε για ειδικά προβλήματα της πατρίδας σας δώστε μας στοιχεία για να δούμε πού έγινε το πρόβλημα, αν είναι δικό μας ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Αλλά θέλουμε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες και καλό θα ήταν να μας τις ε, στείλετε γραπτός. Τώρα, μιλήσατε για το παρατηρητήριο αγοράς γάλακτος. Σίγουρα χρειαζόμαστε έγκαιρα στοιχεία, επίκαιρα και αξιόπιστα για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς γάλακτος. Και αυτό θα βοηθήσει το παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος και σας είπα την τελευταία φορά, εξέτασα το ρόλο του παρατηρητηρίου και πώς θα το διαρθρώσουμε και θα πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε το παρατηρητήριο, πώς θα έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στο παρατηρητήριο αγοράς Γάλακτος και πιο επίκαιρα στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και ιδιαίτερα τις μείωση τιμής γάλακτος, κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τους παραγωγούς. Επίσης χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό άμεσης ε, αντίδραση σε ό,τι αφορά τα στοιχεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει το παρατηρητήριο. Και αν το εφαρμόσουμε, καταφέρουμε και το εφαρμόσουμε και σε άλλα προϊόντα, τόσο το καλύτερο. Γιατί είχαμε καταργήσει, αν έχουμε καταργήσει ποσοστό και ζαχάρο για παράδειγμα, παρόμοιο σύστημα θα μπορούσαμε να είχαμε και για τη ζάχαρη το 2017. Δεν θα αναθεωρηθεί, ε, θα το σύστημα, αλλά θα το εξετάσουμε γιατί αν συνεχίσουν να πέφτουν οι τιμές όπως ε, είπατε και εσείς κύριε Λαπέ και κύριο Νίκολσον, θα πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε τους μηχανισμούς που δίνει η αναθεώρηση για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση. Σε ό,τι αφορά τη χώρα προέλευσης, πρόσφατα εγκρίναμε εκθέσεις, δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη, αλλά η καθυστέρηση οφείλεται στη περίπλοκη διαδικασία που ισχύει και υπάρχει ανάγκη ε, ταυτόχρονης εφαρμογής ε, των εξέσεων και η οικειοθελή σήμανση είναι μια λύση και δίνει την ευκαιρία και στους καταναλωτές ε, να διαλέξουν προϊόντα που έχουν και την, τα στοιχεία προέλευσης. Αυτό προαιρετικά μπορεί να το αναφέρει ο κλάδος και θα δούμε αν χρειαστεί δεσμευτική ε, μνήα της προέλευσης. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα εφαρμοστεί ομοιόμορφα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει η προαιρετική αναφορά της προέλευσης για να δούμε περαιτέρω τι θα γίνει. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της γεωργίας στα πλαίσια της μετανάστευσης και της ε, πολιτικής ασφάλειας, ε, στενίζομαι πλήρως αυτά που είπατε, κύριε Νέκοφ, για το θέμα αυτό και η μεταφορά της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Αφρική, γιατί οι αφρικανικές χώρες χρειάζονται αυτές τις γνώσεις, τεχνογνωσία, για να μπορέσουν και οι χώρες Αφρικής να παραγάγουν τα δικά τους προϊόντα και να μειωθεί και η μετανάστευση. Βέβαια, και η Γεωργία θα διδραματίσει ρόλο, αλλά δεν θα είναι μόνο ο δικό τη ο ρόλο. Χρειαζόμαστε και μέσω και μακροπρόθεσμε λύσει. Και η πολιτική πιστιστική ασφάλεια επίση είναι σημαντική. Και προσπαθούμε με την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη να προωθήσουμε τα σωστά μηνύματα για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν η γεωργία και η πιστιστική ασφάλεια ε, στη μετανάστευση και στη γεωργική πολιτική. Βαλτικές χώρες. Δεν διάβασα ακόμη το έγγραφο της ε, Λιθουανίας για τις προτάσεις ε, βελτίωσης της κατάστασης. Θα δούμε. Θα το κοιτάξω και θα δω αν μπορούν να εφαρμοστούν και να είναι αποτελεσματικές. Είναι μείζον το πρόβλημα και που δεν, είναι, δεν το υποτιμώ στις βαλτικές χώρες ειδικά Γι' αυτό ακριβώ πέρυσι αντιδράσαμε στο γαλακτοκομικό τομέα και παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυ. Όντω η τιμή που αναφέρεται είναι ανησυχητικά χαμηλή. Και περιμένω τι ιδέε τη ε, Λιθουανία για να βοηθήσουμε τι βαλτικέ χώρε. Ο κύριο Ρεμπέκα, που είναι από τη Ρουμανία, μίλησε για εξάμεινη παράταση του προγράμματο αγροτική ανάπτυξη. Προ το παρόν δεν, σας, δεν μπορώ να σα δώσω το πράσινο φω, γιατί δεν είναι ε, μόνο η δική μου υπηρεσία. Έχουμε και άλλες διευθύνσεις ε, που είναι συνορμόδιες και που διαφωνούν με την παράταση. Πάντως προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ικανότητα απορρόφησης ε, των προγραμμάτων για το πρόγραμμα 2013-2017 και να θελήσουμε τη γραπτή διαδικασία σε ό,τι αφορά την αύξηση σε ορισμένου τομεί από 3 σε 5%. Οπότε αυτό θα απαντήσουμε στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία που επίσης είχε πρόβλημα με την απορρόφηση. Η Ελλάδα επίσης έχει πρόβλημα χαμηλής απορρόφησης. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις αρχές και να βελτιώσουμε την εφαρμογή του προηγούμενου σχεδίου για να μπορέσετε να εκταμιεύσετε περισσότερα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των νέων γεωργών, νομίζω ότι ε, εσείς ε, διαγράφοντας το 25% το ανώτατο όριο για την ΚΑΠ είχατε πολλά καλά μέτρα. Ε, εμείς προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την ΕΤΕ για χαμηλό το καδάνια και να μπορούν οι νέοι γεωργοί να έχουν πρόσβαση στο δανεισμό για να μπορέσουν να αναλάβουν και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Πάντως το πρόγραμμα με την ΕΤΕ θα πρέπει να ενταχθεί στο δικό σας πρόγραμμα ανάπτυξη πέθρου. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου ε, ένα καθεστώς ε, εγγυήσεων για τους ε, νέους γεωργούς. Ο κύριος Χαϊτεμα αναφέρθηκε σε θέματα που εκπίπτουν των αρμοδιοτήτων μου. Πάντως ε, τα σημείωσα και θα τα διαβιβάσω στον Επίτροπο Κάιτες, που είναι ο αρμόδιος Επίτροπος Υγείας, σε ό,τι αφορά την γεωργία και την κτηνοτροφία, την καλλιέργεια φυτών και την εκτροφή ζώων. Το Φεβρουάριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε εξυγχρονισμό των κανόνων ζωοτεχνικής. Αλλά επαναλαμβάνω, ο αρμόδιος ε, επίτροπος είναι ο κ. Ε, και θα του ζητήσω να σας στείλει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Μα ανησυχεί και το φαινόμενο τη μικροβιακή αντίσταση, που βέβαια δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά παγκόσμιο από το 2001 προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μικροβιακή αντίσταση με πρόληψη, έρευνα, ανάπτυξη προϊόντων, διεθνή συνεργασία και παρακολούθηση. Και μάλιστα έχουμε παρατείνει την περίοδο μέχρι το 2015 και έχει προγραμματιστεί και μία αξιολόγηση για φέτο για τι στρατηγικέ δράσει του σχεδίου δράση για να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντίσταση. Σε ό,τι αφορά την ε, ευημερία των ζώων, έχουμε πλήρη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις υψηλότερες παγκοσμίω προδιαγραφές για το θέμα της ευημερίας των ζώων. Πρέπει να εφαρμοστούν όμως τα μέτρα. Τώρα προτεραιότητα είναι η εναρμόνιση, αλλά αυτό αφορά τα κράτη-μέλη. Βλέπω ότι αρχίζετε και δυσανασχετείτε. Θα ολοκληρώσω εντός ολίγου οι ορεινέ περιοχές, οι εξόχω απόκεντρε περιοχές είναι θέμα των κρατών μελών. Και η ερώτηση του, Νταντάν, ε, του κ. Νταντάν, υποβάλαμε αίτηση για άρση του ρωσικού εμπάργου. Μα συνεχώς προσπαθούμε να, ε, να επισημάνω αυτό το πρόγραμμα ε, το πρόβλημα στους Ρώσους που ζητούμε να αποσυρθούν, αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ουκρανία και αυτό εντάσσεται στη γενική πολιτική ασφάλεια. Και βέβαια η Γεωργία υφίσταται τις ε, συνέπειες αυτής της πίεσης γιατί χρησιμοποίησε τη Γεωργία και το εμπάργο Ρωσία ως αντιπερισπασμό στα αιτήματά μας για την Ουκρανία. Πάντως με την κυρία Μοκαρίνη προσπαθούμε να ε, ε, πείσουμε τους Ρώσους να λογικευτούν. Οπότε σας διαβεβαιώ κύριε Νταντάν, δεν ξεχνάω καθόλου το θέμα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη συνεργασία, τη συζήτηση και προσβλέπω και στη συνέχιση τη συνεργασία στο μέλλον. Ό,τι δεν απάντησα απευθείας θα σας στείλω γραπτός απαντήσεις. Ευχαριστώ. Έχω μια καταπληκτική είδηση να σας ανακοινώσω. Μέσα σε μια μισή εβδομάδα θα τα ξαναπούμε με τον Επίτροπο στις 8 Ιουνίου συγκεκριμένα, στο Στρασβούργο, στις 7 το απόγευμα. Θα μιλήσουμε για την ανταγωνιστικότητα. Εκεί θα ακούσουμε και πάλι τον Επίτροπο και την αρμόδια Επίτροπο Ανταγωνιστικότητας. Τον αρμόδιο Επίτροπο Ανταγωνιστικότητας, την αρμόδια Επίτροπο την κυρία Βεστάγκεν. Οπότε στις 8 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, το απόγευμα 7 η ώρα, σημειώστε στις ατζέντες σας και θα ψηφίσουμε και την έκθεση Νίκολσον εκεί για το γάλα. Οπότε θα ξαναέχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, προσβλέπουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Πολύ χρήσιμη ήταν η σημερινή. Και επίσης περιμένω τις προτάσεις σας και να εγκρίνουμε και τις συστάσεις των συντονιστών. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Εγκρίνονται οι συστάσεις των συντονιστών. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς λέει ο Πρόεδρος, γιατί μας επιτρέψετε να ακούσουμε μέχρι τέλος τις απαντήσεις του Επιτρόπου που ήταν πολύ σημαντικές. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλή επάνωδο στις πατρίδες σας.